Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, μάλλον καθίστε. We will start our meeting, please. Thank you very much. Λοιπόν, ξεκινάμε την ε, απόψινή μας συνεδρίαση. Θα μελετήσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία αρχικά και ιδίω θα συζητήσουμε την περίπτωση του κύριου Ανταργατσέφ Τσέγκε. Είχε πάει μια αντιπροσωπεία της υποεπιτροπής μας στην Αιθιοπία τον Ιούλιο του 2013. Είχαμε επισκεφθεί και την Αφρικανική Ένωση και τις Αιθιοπικές Αρχές και αυτή η ενημέρωση έρχεται σε συνέχεια αυτής της επίσκεψης. Στο μεταξύ έχουν προκύψει ανησυχητικά γεγονότα, άκρως ανησυχητικά θα τα χαρακτήριζα, διότι συνελήφθη ε, με πάρα πολύ περίεργο, παράδοξο τρόπο ο κύριος Τσέγκη και κρατείται και δεν είναι ο μόνος. Πολλοί bloggers από την Zone 9, τη Zone 9 αυτό το blog και είμαστε εδώ για να αναλύσουμε αυτή την κατάσταση όσοι γνωρίζουν ε, την υπόθεση αυτή. Βέβαια έχουμε και την εκπρόσωπο της Πρεσβείας της Αιθιοπίας, εκπροσώπους της Κομισιόν του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δούμε ποια είναι η κατάσταση και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί στόχος της υποεπιτροπής μας είναι η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία μάλλον η, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Εγώ άκουσα όλες τις ε, πληροφορίες που κάνουν λόγο για την μεγάλη βελτίωση της ε, κατάστασης στην Αιθιοπία. Οδεύει στο δημοκρατικό μονοπάτι τα τελευταία 30 χρόνια, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Οικονομικά επίσης έχει αναπτυχθεί, κατά καταπολεμάει και τη φτώχεια. Αυτά τα συζήτησα με τον πρέσβη. Και βέβαια συζητήσαμε ότι δεν υπάρχει σειρά πρώτα οικονομική ανάπτυξη, μετά εκδημοκρατισμό και μετά ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά πρέπει να πηγαίνουν όλα μαζί παράλληλα. Και ο πρέσβη συμφώνησε απόλυτα και είναι και στη διάθεσή μα. Υπάρχει εκπρόσωπο τη πρεσβεία εδώ. Θα συλλέξει όλε τι πληροφορίε και θα μα ενημερώσει από την πλευρά του. Υπάρχουν διάφοροι συμμετέχοντε στο πάνελ. Καταρχά η κυρία Φώα, ε, στρατηγική διευθύντρια τη ομάδας Ανατική Ποινή από την ε, μη κυβερνητική οργάνωση ρεπρί που όπω γνωρίζετε επεξεργάζεται όλα αυτά τα θέματα με μεγάλη αποτελεσματικότητα και θα σας δώσω κυρία Φώα για πέντε λεπτά το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση. Ε, εγώ εργάζομαι για αυτή την υπόθεση εδώ και αρκετούς μήνες, τρεις για την ακρίβεια, από τότε που απήχθη στην Ιεμένη τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Ο Αντεγάτου Τσέγκε είναι Βρετανός υπήκος, ο οποίος έμενε στο Λονδίνο με την ε, ε, συμβία του και δύο παιδιά ε, απήχθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ανάτης Εμένης Ιεμένης ταξίδευε από τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς την Ερυθρέα απόλυτα νόμιμα δεν γνωρίζαμε που η οικογένεια μάλλον δεν γνώριζε, ούτε η Βρετανική κυβέρνηση δεν γνώριζαν για δύο εβδομάδες που βρισκόταν μέχρι ότου στις 7 Ιουλίου η Αιθιοπιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ήταν υπό τη δική τους ε, ε, φρουρά εφού είχε μπει στο, σε ένα αεροπλάνο και είχε προσγειωθεί στην Ερυθρέα την ημέρα που απήχθη. Και πιστεύουμε όλα αυτά βέβαια με ε, παραβίαση το κάθε διεθνού νομοθεσίας. Από τότε κρατείται σε κάποια τοποθεσία που η, κυβέρνηση της Αιθιοπίας δεν έχει αποκαλύψει στη Βρετανική κυβέρνηση, ούτε στην οικογένεια του Ανδεγάτσου. Είχε μια σύντομη συνάντηση με έναν πρέσβη, αλλά διαρκώς ε, δεν του δίνεται πρόσβαση στις προξενικές αρχές, ούτε δικαίωμα να φύγει από τη χώρα, ούτε ανεξάρτητη ιατρική ε, βοήθεια. Αυτή τη στιγμή είναι, είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Ε, η απόφαση αυτή λήφθη τη απουσία του ερήμην του το 2009 και έχουμε πολύ μεγάλες εμφωλίες όσον αφορά τη δικαιοσύνη αυτής της δίκης. Ε, η κυβέρνηση τη Ιωπία δεν έχει δώσει καμία διασφάλιση ότι δεν θα εκτελέσει την ποινή παρά τα αιτήματα των Βρετανών και άλλων οργανώσεων. Εμείς και η οικογένειά του βεβαίω ανησυχούμε πάρα πολύ για την υγεία του και για την ε, κακομεταχείριση στη διάρκεια της κρατησή του γιατί χρησιμοποιείται η βία και τα βασανιστήρια κατά των πολιτικών κρατούμενων. Τον Ιούλιο είδαμε δύο ε, βίντεο στην ε, τηλεόραση της Αιθιοπίας ε, με ανακρίσεις του Αντεγκάτσου. Οι Βρετανοί εμπειρογνώμονες εξέτασαν τα, τις ταινίες αυτές και η Βρετανός ψυχίατρος είπε ότι είχε σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ψυχική του υγεία τα τραύματα που μπορεί κανείς να έχει μετά από κράτηση και βασανιστήρια ε, μπορεί να είναι πολύ σοβαρά. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί ε, στη διάρκεια της κράτησής του και δεν το ξέρουμε γιατί δεν μας έχει δοθεί καμία πρόσβαση. Ε, είναι θύμα απαγωγής, παράνομης κράτησης και πιθανότατα βασανιστήριων. Όπως σας είπα, είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Η καταδίκη του έγινε ερήμην. Η Βρετανική κυβέρνηση απαιτεί να απελευθερωθεί και να επιστραφεί στην οικογένειά του, ε, επιγόντως μάλιστα. Όπως σας είπα όμως, η Αιθιοπία αρνείται να αναγνωρίσει ότι έχουν ε, γίνει εγκλήματα κατά του συγκεκριμένου ατόμου, αρνείται να αναγνωρίσει ότι έχουν παραβιαστεί τα βασικά του δικαιώματα υπό το διεθνέ Δίκαιο, το δικαίωμα πρόσβαση νομική εκπροσώπηση το δικαίωμα σε ανεξάρτητη ιατρική περίθαλψη. Είναι τελείω αδύναμο. κρατείται σε άγνωστο μέρο, ε, εδώ και πάνω από τρει μήνε. Η οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ιδέα που βρίσκεται, ούτε πώ είναι η ψυχική του ή η σωματική του υγεία. Υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με το γιατί απήχθηκε, γιατί τώρα κρατείται στην Αιθιοπία, ήταν και είναι ε, ηγετικό στέλεχος ε, το Τζιμ Λεφτά που είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης αρκετά ισχυρό στην Αιθιοπία ε, έχουν συλληφθεί πολλοί πολιτικοί ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί. Ε, έχει, γενικά ασκείται μεγάλη πολιτική καταστολή από το καθεστώς της Αιθιοπίας και έχει επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία πριν από τις εκλογές που προβλέπονται για το 2015 ε, πρόσφατα ο ειδικό απεσταλμένος του ΙΕΕ και του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων κτλ ότι υπάρχουν για την ισχύουσα κατάσταση στην ε, Αιθιοπία και κάλεσαν την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να απελευθερώσουν όλους τους ανθρώπους που αυθαίρετα κρατούνται υπό την, ε, ε, με, την δικαιολογία της, της τρομοκρατίας. Θέλουν λοιπόν να αφήσουν στου, τους πολιτικούς αντιπάλους τους και τους θρησκευτικού αντιπάλους να ασκούν τα δικαιώματά τους χωρίς εκφοβισμό η ε, η Αιθιοπία επικρίνεται βεβαίως ε, και πολλοί από τους ε, κρατούμενους αυτούς έχουν καταδικαστεί, έχουν εκτελεστεί και δεν τους έχει δοθεί καμία, κανένα δικαίωμα για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους ή να παρουσιάσουν αποδείξεις για να ενάντια στις κατηγορίες που τους έχουν απευθυνθεί. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα απελευθερωθεί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε λάβει τη δήλωση, το statement ε, της Βρετανικής κυβέρνησης. Νομίζω το μοιράσαμε και πρέπει να το έχετε στη, στα έδρανά σας. Εκεί λοιπόν ε, επιβεβαιώνει η Βρετανική κυβέρνηση τα λόγια της κυρίας Φώα. και εκφράζει τη λύπη της και καταγγέλει το γεγονός ότι δεν έχει πρόσβαση στον κρατούμενο. Περιγράφει το πώς έγινε αυτή η σύλληψη, περί, ουσιαστικά πρόκειται περί έκδοσης. Έχετε το σχετικό κείμενο στα έδρανά σας. Η κυρία Γκόμες νομίζω Ζήτησε το λόγο, αλλά δεν ξέρω. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το σημείο ή να ακούσουμε πρώτα και ο κύριο Χόιτ. Ή περιμέ... να περιμένουμε καλύτερα πρώτα να ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Κύριε Χόιτ, θέλετε το λόγο. Νομίζω ότι η παρουσίαση αυτή είναι πολύ σημαντική και είμαι πολύ ευγνώμων. Ε, ως Βρετανός σας χαιρετίζω και θέλουμε να Ξέρετε ότι έχουμε λάβει τη δήλωση του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και ε, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος της συζήτησης θα σας υποστηρίξουμε ε, πλήρως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώ, ε, το, το να πω το οτιδήποτε άλλο μάλλον δεν θα προσθέσει τίποτα σε αυτά που είπατε εσεί ήδη. Απλά ήθελα να ξέρετε ότι σα ακούμε και ότι υποστηρίζουμε πλήρω την θέση της και νομίζω, Πρόεδρε, ότι και εσείς θα καταλήξετε στο ίδιο συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Έμα Κίλη, επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Frontline Defenders. Θα μας μιλήσει για την κατάσταση των bloggers ε, της Zone 9, zone 9. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση του Frontline Defenders. Η Frontline είναι μια οργάνωση που σκοπός είναι να παράσχει γρήγορη δράση για να ε, προστατεύσει ακτιβιστές ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των ε, κατηγορουμένων και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση 9. Στις 17 ε, Ιουλίου οι εθοπικές αρχές κατηγόρησαν 10 ε, ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία του 2009. 7 από αυτούς είναι μέλη του Ζώνη 9, ενώ τρεις άλλοι είναι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι. Βρίσκονται καταδικασμένοι, είναι στη φυλακή και στι 15 Οκτωβρίου αναμένεται η δίκη του. Η Ζώνη 9 είναι μια ομάδα blogger που ε, συζητούν ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντα στην Αιθιοπία. Μα ανησυχεί το γεγονό ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο και έχει επιχειρηθεί να σιωπήσουν όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τους. Πιστεύουμε μετά από ανάλυση της κατάστασης και των κατηγοριών ότι οι αρχές σκοπίμως χρησιμοποιούν στιμένες κατηγορίες όπως ε, ε, οι διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Jimbot 7 και με το Roman Liberation Front Επίσης, ε, κατηγορίες για αποσταθεροποίηση του έθνους, που κατηγορίες που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και τη θανατική καταδίκη. Ως ένδειξη χρησιμοποιείται επίσης και η χρήση από την πλευρά των blogger του Security in a Box, το οποίο είναι ε, διαθέσιμο στο ίντερνετ. Πρόκειται ε, για ένα λογισμικό που ε, δίνει τη δυνατότητα στους ακτιβιστές αυτούς να ε, επικοινωνούν ασφαλώς, με ασφάλεια στο ίντερνετ. Το περιεχόμενο αυτού του software είναι δωρεάν, είναι διαθέσιμο και νόμιμο. Οι αρχές της ε, υπονοούν ότι ε, η χρήση αυτού του software είναι απόδειξη, είναι ένδειξη μάλλον ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλαν ε, απλά και μόνο χρησιμοποιώντας το software να ε, χρησιμοποιήσουν βία. Στην Αιθιοπία λοιπόν η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. υπάρχουν περιορισμοί της ελευθερίας, του λόγου, της συνάθρησης, υπάρχουν αυθαίρετες συλλήψεις η κατασταλτική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ήταν επιτυχημένη. Πολλοί ε, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι έχουν ε, αναγκαστεί να φύγουν ε, από τη χώρα από φόβο. Από τότε που εκφράστηκαν αυτές οι κατηγορίες, οι πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι έχουν λάβει άμεσες και πολλοί έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη, χώρη, τη χώρα. Τον Αύγουστο μόνο 14 δημοσιογράφοι από γνωστά ΜΜΕ έχουν ζητήσει άσυλο στην Κένια. Η Αιθιοπία επίσης επιβάλλει ε, πολλούς περιορισμούς στο ίντερνετ και στις ψηφιακές επικοινωνίες. Είναι η μοναδική χώρα της υποσαχάριας Αφρικής που φιλτράρει, ε, σύμφωνα με το Freedom House, τις επικοινωνίες. Επίσης υπάρχει ε, από το Open Network ε, μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι η αιθιοπική κυβέρνηση επιβάλλει φιλτράρισμα ε, στο διαδίκτυο. Επίσης, ε, πολλές φορές τίθεται στο στόχαστρο πολιτικό περιεχόμενο και συγκεκριμένα blogger και μάλιστα δίνονται οδηγίες για να κατεβάσουν ε, περιεχόμενο από το ίντερνετ, ακόμη και σελίδες στο facebook. Γίνονται υποκλοπές ε, και το software που χρησιμοποιούν οι αρχές είναι ε, εξαιρετικά προηγμένο με τη βοήθεια της κινέζικης κυβέρνησης. Κατά συνέπεια λοιπόν η Frontline χαιρετίζει το, την, ε, την δήλωση που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και επίσης χαιρετίζουμε και τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 30 Ιουλίου όπου οι ε, πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις σε σχέση με τους blogger και ζητούν από τις αρχές της ε, οι δίκες να διεξαχθούν με βάση τα διεθνή πρότυπα να έχουν οι κατηγορούμενοι δικαίωμα επικοινωνίας με δικηγόρους και με τις οικογένειές τους και να διεξαχθούν δίκες χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Οπότε θα θέλαμε να ε, αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται ε, για να ρωτήσουμε τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα δώσω ακριβώς το λόγο στην κυρία Γκαρθία Γκυγέν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που είναι υπεύθυνα για τη Αιθιοπία. Ναι, ευχαριστώ, αλλά καλύτερα να δώσω το λόγο στον ε, προϊστάμενό μου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Λέγομαι Ντίτμαρ Κρίσλερ και είμαι ο αναπληρωτής διευθυντής ε, του τμήματος ε, της ΕΙΕΤ που ασχολείται με την Ανατολική Αφρική. Κύριε Πρόεδρε, εμείς παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία και τον τελευταίο μήνα πράγματι βιώσαμε ανησυχητικές εξελίξεις, παίξαμε μάρτυρες ε, ε, συλλήψεων bloggers, δημοσιογράφων, μελών ε, της αιθιοπικής αντιπολίτευσης, τα είπε και η ΕΜΑ μόλις πριν. Η κατάσταση απαιτεί την προσοχή μας, ιδίως στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών που θα λάβουν χώρα τον επόμενο Μάιο στην Αιθιοπία. Η Ευρωπαϊκή η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αμπέμπα παρακολουθεί από πολύ κοντά τα όλα γεγονότα, τις εξελίξεις αυτές και ιδίως ε, τη δίκη ε, ή τις δίκες ε, που θα διεξαχθούν μετά από τις συλλήψεις αυτές. Έχουμε επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη δημιουργίας χώρου για έναν γνήσιο πολιτικό διάλογο στην Αιθιοπία για να είναι εγγυημένη η ελευθερία έκφρασης ε, και συνάθρησης, ε, συνεταιρίζεστε. Έχουμε πολλές ανησυχίες σε ό,τι αφορά ε, αυτό το Anti-Terrorist Proclamation. Γιατί με αυτή και άλλες δραστηριότητες περιορίζονται, περιορίζεται η ελευθερία των bloggers, των δημοσιογράφων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει δημοσιεύσει μια δήλωση, συγκεκριμένα 6 Μαΐου, η ημερομηνία που δημοσιεύθηκε και καλούμε τις αρχές ε, να βεβαιωθούν στην περίπτωση των ε, συλληφθέντων bloggers και δημοσιογράφων ε, θα γίνουν οι δίκες με βάση το αιθιοπικό δίκαιο και σε σεβασμό προς τα διεθνή πρότυπα και κανόνες. Επιπλέον, και είμαι γνώμη προς την ΕΜΑ γιατί ανέφερε και η ίδια ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αντισαμπέμπα στις 30 Ιουλίου εξέδωσε και αυτή μια ανακοίνωση εκφράζοντας ε, την ε, ανησυχία της για τις συλλήψεις μελών ε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτά τα θέματα, κυρία Πρόεδρε, τα θέτουμε συνεχώς στις αιθιοπικές αρχές, στο πλαίσιο του διαλόγου άρθρο 8 που έχουμε την αιθιοπική κυβέρνηση και στο υψηλότερο επίπεδο, γιατί τακτά συναντώμεθα με τις αρχές ε, της Αιθιοπία και εδώ και στην Αντισαμπέμπα και συζητούμε μαζί τους όλα τα ζητήματα που μας ανησυχούν. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω ότι εκτός από τις διπλωματικές μας δραστηριότητες ε, συνεργαζόμαστε και προς ε, τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αιθιοπία μέσω στοχευμένης αναπτυξιακής βοήθειας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο 11ο ενδεικτικό πρόγραμμα ε, του ΕΤΑ για την Αιθιοπία έχουμε λάβει 52 εκατομμύρια ευρώ για την χρηστή διακυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών. Και στόχο ε, των κονδυλίων αυτών είναι να ενισχυθεί η διαδικασία του εκδημοκρατισμού στην Αιθιοπία. Τέλο, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Ανταργκάτσεφ, παρακολουθούμε ε, την κατάσταση σε στενή συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές. Έχουμε παράσχει την βοήθειά μας, ε, την υποστήριξή μας και νομίζω ότι η βασική ανησυχία έγκυται στο κατά πόσον θα υπάρξει μια νόμιμη ε, δίκη και διαδικασία, ιδίω πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσον ήταν νόμιμη η έκδοσή του στην Αιθιοπία, η προσαγωγή του, η σύλληψή του και επίσης η κατά πόσο του παρασχέθηκε προξενική υποστήριξη και νομική υποστήριξη. Φυσικά είμαστε κατάφορα αντίθετοι στα αντική ποινή που φαίνεται ότι το έχει επιβληθεί. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ε, κατάσταση στην Αιθιοπία. Θα συνεχίσουμε άμεσα στις αιθιοπικές αρχές ε, να εκφράζουμε τις ανησυχίες μας και δημοσία βέβαια θα αντιδράσουμε εφόσον απαιτηθεί από τις εξελίξεις κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. κατάλαβα καλά, είστε ο αρμόδιος για την Αφρική, είπατε. Είναι ο αναπληρωτής τομέας για την, για την Ανατολική Αφρική. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας, και αυτό θέλω να κάνω, θα προτιμούσα να είχατε εμβαθύνει λίγο παραπάνω πάνω στο τι, ε, ποια θα είναι η δράση, ποιες θα ενέργειες, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Λέτε αν απαιτηθεί από τις περιστάσεις θα παρέμβετε, θα αντιδράσετε. Εγώ νομίζω ότι απαιτείτε τις περιστάσεις να αντιδράσετε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αναγκόμης, προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, κάπως την ξέρω την Αιθιοπία. Ήμουν εκεί το 2005, επικεφαλής της ε, αποστολής παρατήρησης εκλογών. Κάποιες φορές το χρησιμοποιεί αυτό η Αιθιοπία σε επιχείρημα ε, για να ουσιαστικά να με συκοφαντήσει, να με δυσφημίσει, γιατί εγώ το μόνο που έκανα όμως είναι να είμαι αντικειμενική και να λέω την αλήθεια. Είμαστε 200 παρατηρητές εκεί και εγώ είπα πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ενώ υπήρχε προσέλευση μαζική της κάλπες, πίστευαν δηλαδή σε εκλογές οι Αιθίωπες, τα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση των ψήφων ήταν νοθευμένα σε βαθμό που ε, να προσανατολίζονται εντελώς. Παρ' όλα αυτά και παρότι προσπάθησαν να τα καλύψουν με την καταμέτρηση πήγαν 24 στην αντιπολίτευση. Έκτοτε, επαναλαμβάνω, ε, προσπαθούν να μειώσουν ε, τις δηλώσεις μου στην Αιθιοπία. Εγώ όμως έχω συναντήσει διαφόρους ε, στην Αιθιοπία. Συνάντησα και τον κύριο Τσέγκη. Τον συνάντησα και αφού τον είχαν τότε στη φυλακή και πολλοί άλλοι αντιπολίτευσεις ήταν στη φυλακή τότε για 1,5 χρόνο. Μετά κατάφερε να πάει στην Βρετανία και είχα επαφή μαζί του και με πολλούς άλλους από την Εθνική Διασπορά. Και φυσικά χαίρομαι ε, για αυτά που είπατε. Δεν θέλω και εγώ να πω ότι ουσιαστικά πρόκειται για παράδοση ενός ανθρώπου από την Ερυθρέα στην Αιθιοπία. Είναι τραγική η κατάσταση. Ένας άνθρωπος όμως που είναι Βρετανός. Έχει καταδικαστεί επίσης σε θάνατο και φοβούμε. Φοβούμε για τη ζωή του. και αν έχει σωθεί μέχρι τώρα η ζωή του, αυτό οφείλεται στην αντίδραση τη διεθνού κοινότητα. Ακόμη και το Foreign Office αναγκάστηκε δημοσία να εκφραστεί, γιατί ξέρω ότι έχει του πληροφοριοδότες του και του συμβούλου του στην Αιθιοπική Κυβέρνηση, το Foreign Office και κάποιου του γνωρίζω μάλιστα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η παράδοση θα μπορούσε να είχε γίνει αν δεν ήξεραν, αν δεν είχαν πλήρη γνώση οι Βρετανοί γι' αυτό. Πάντως, ε, μετά από όλα όσα υπόθηκαν, ε, ε, εξακολουθεί η ανησυχία μου για τον κύριο Τσέγκη να είναι μεγάλη. Είναι ανυπόφορη αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανική κυβέρνηση έχουν την υποχρέωση να κάνουν πολύ περισσότερα από το να εκδίδουν απλά κάποιες δηλώσεις και ανακοινώσει. Και ακόμη και στι συζητήσει που γίνονται στην Αιθιοπία, υπάρχει μεγάλη, μεγάλος μεγάλη επιφυλακτικότητα. Σίγουρα είναι μια χώρα σημαντική για την όλη περιοχή, που είναι ένας μείζον εταίρος ε, στη περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού, αλλά θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Πώς θα την κάνουμε τη διαφορά. Δυστυχώς κάποια κράτη-μέλη δεν το θέλουν αυτό. Θέλουν να συνεχίσουν business as usual. μήπως να συνεχίσουν να πολλούν τα φίλτρα για το μπλοκάρισμα των ε, σελίδων ε, των blogs. Όταν είχαμε πάει με την κοινή ε, αντιπροσωπεία, την κοινή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία ΑΚΕ, Ε, ευτυχώς μπόρεσα να πάω και εγώ και είχα πολύ καλές επαφές και με μέλη της κυβέρνησης και μου ζήτησαν να δώσω κάποια μηνύματα προς την αντιπολίτευση εν ώψη της προετοιμασίας των εκλογών του Μαΐου και το έκανα. Του είπα όμως και πολύ ξεκάθαρα, στις αρχές δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να έρθει από την Αλγαπή η αντιπολίτευση εάν δεν είναι αν δεν πληρούνται οι βασικές αρχές για τη δημοκρατία, για δίκες εκλογές, με την καταστολή που όλο και χειρότερη γίνεται στους bloggers, στους δημοσιογράφους, στους ε, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί η κατάσταση και ελπίζω να έχουμε μια άλλη αντίδραση. Ξέρετε ότι μετά το 2005 στάλει μια άλλη αποστολή παρατήρηση ε, εκεί και δεν μπόρεσε καν να εκπονήσει ή να δημοσιεύσει την έκθεσή τη. Ένα Ολλανδό άλλο να θυμάμαι καλά. Ο Τέι, Τέι Μπέρμαν. Δεν πρέπει να συνεχιστεί, ούτε να επαναληφθεί. Γιατί ξέρετε ότι όταν ήμασταν εκεί, είχαμε τον κύριο Σκίντερ Νέγκα, έναν δημοσιογράφο που μα ανησύχει ιδιαίτερη περίπτωσή του, που είχε βραβευτεί στις και ένας δεύτερος ε, καρκινοπαθής ε, δημοσιογράφος. Πήγαν οι συμπρόεδροι, ο Λουί Μισελ και κάποιος άλλος και επισκέφθηκαν στις φυλακές. Αλλά τι τους δείξαν εκεί. Τις εγκαταστάσεις, τις φυλακής του που είναι η Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ, επικεφαλή αντιπροσωπεία που πήγε πέρυσι, δεν μπόρεσε να, το 12 μάλλον, δεν μπόρεσε να πάει σε αυτή τη φυλακή. Τέλο πάντων, όταν οι συμπρόεδροι αυτή τη κοινή αντιπροσωπεία ε, και πήγαν εκεί, μετά είπαν ότι όλα ήταν πολύ καλά, μέχρι και πρόσβαση στο ίντερνετ λέει είχαν κρατούμενοι. Και δεν είχαμε εμεί πρόσβαση στο ίντερνετ. Αλήθεια. Πώ μπορεί αυτοί του οποίου κατηγορούν για τρομοκράτε να έχουν πρόσβαση στη φυλακή, στο ίντερνετ και εμεί στα ξενοδοχεία μα να μην έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει τεράστια ευθύνη. Έχει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή. Και έχουν ε, και η μεγάλη ευθύνη που δεν αντέδρασαν με αποφασιστικότητα απέναντι στη χώρα με την οποία έχουν σχέσει. Πρέπει να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Αιθιοπία στο πλαίσιο των συμφωνών Κοτονού. Εγώ τα είπα και τα ξανάπα και τότε με την αντιπροσωπεία και είχα ρωτήσει και τον ε, Επίτροπο Πίμπαλξ και τον, ε, νομίζω ήταν πρωθυπουργό της Λιθουανίας εκπρόσωπος του Συμβουλίου και ήταν και παρόν ένας εκπρόσωπος της Αιθιοπίας, της κυβέρνησης τη Αιθιοπίας που έλεγε δεν υπάρχουν ε, πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές της Αιθιοπίας, μόνο τρομοκράτες. Ούτε ο κύριος Πίμπαξ, ούτε ο δεν ξέρω ποιος, κύριος Βιτσιούτε ή κάτι τέτοιο από τη Λιθουανία είχαν την ειλικρίνεια και την αξιοπρέπεια να πούν παρά όλε αυτέ τι δηλώσει που γίνονται χωρί κανένα αποτέλεσμα, ότι όχι, υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι στην Αιθιοπία. Και ότι δεν πληρώνει τι υποχρεώσει του πλαίσιο των συμφωνών με η Αιθιοπία. Ana εγώ με σου dar την στην κυρία Φώα με Μου ζήτησε η κυρία Φώα το λόγο, λέει πρόεδρο. Θα, θα, θα της τον δώσω. Σα ευχαριστώ και πάλι. Να συνεχίσω από κάτι που είπε η Άννα Γκόμες και να ρωτήσω τον κύριο Χάουετ για τη Βρετανική θέση. Γιατί ενώ έχουν κάνει δήλωση και μάλιστα αρκετά στεναρή σε σχέση με τη πιθανή κακομεταχείριση για την παράνομη έκδοση του κυρίου Τσέγκε, από όσο γνωρίζω δεν ζητούν άμεση και ανεφόρον απελευθέρωσή του που είναι το μήνυμο κατά τη γνώμη μου που θα έπρεπε να ζητούν, δηλαδή προξενική πρόσβαση και η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε σε αυτό, ότι σχεδόν στην ουσία αγνοούν τους, μάλλον δεν κάνουν τίποτα. Μία προξενική επίσκεψη μόνο στους Αιθίωπες και πραγματικά δεν ε, είναι έτσι ε, έντονη ανταπόκριση του. Έχω εδώ μια επιστολή που έλαβα από την κυβέρνηση που αναγνωρίζει ότι οι προηγούμενε καταδίκε έγιναν ερήμην και ε, προκαλούν διάφορε ανησυχίε. εγιναν ερημην και προκαλουν διαφορε ανησυχιε κρατειτε με κάθε παράβαση, ε, με παράβαση μάλλον κάθε διεθνού νομοθεσία και η Βρετανική κυβέρνηση δεν ζητά την απελευθέρωσή του. Απήχθη, ε, τον έδεσαν, τον ε, ρίξαν μέσα σε ένα αεροπλάνο. Είναι ένα Βρετανό υπήκο που πάει από τη μια μέρα, ένα μέρο στο άλλο. Ξέρετε πολύ καλά τη χώρα, έχετε επιρροή εκεί. Πέρα από τη βοήθεια που μας δίνει, νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ε, και με την ποινική δικαιοσύνη και το πρόγραμμα μας που χρηματοδοτεί η Βρετανική κυβέρνηση στην Αιθιοπία. Έχει να κάνει με εγκληματίες, με ποινικού κρατούμενους και με ε, πολιτικούς κρατούμενους. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς επηρεάζει η Βρετανική κυβέρνηση για το καλό. Ναι, η συζήτηση είναι λίγο μεταξύ μας, αλλά ευχαριστώ για τη γενεδορία σας, Πρόεδρε, και που μου επιτρέπετε. Είναι για καλό σκοπό, είναι δίκαιο το σχολείο σας, νομίζω, και... Τα όσα είπε και η συνάδελφος και φίλοι Γκόμες δείχνουν ότι όλα αυτά ήταν παράνομα Και αυτό είναι ένα σαφέ επιχείρημα σε σχέση με τα όσα ζητάτε, φαντάζομαι και η πρόεδρο θα συμφωνήσει ότι θα μπορούσαμε να πιέσουμε για να αφαιθεί. Εφόσον είναι παράνομα κρατείται, δεν υπάρχει κανένας και νόμιμος λόγος για να παρατείνεται η κράτησή του. Ε, εάν λοιπόν συμφωνείτε να στείλουμε επιστολή στου Αιθίωπες αλλά και στους Βρετανού. Και ελπίζω να έχουμε ίσως μια ευκαιρία να συναντηθούμε και κατηδίαν για να, πούμε, να δούμε πώς θα το συντάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άστρε Βίσιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, λάβαμε κάποιες επιστολές και δηλώσεις που έγιναν στα τέλη Ιουλίου. Ε, δύο μήνες έχουν περάσει έκτοτε. Μπορεί κανείς να μας πει ενδιάμεσα τι διαβήματα έγιναν. Μεταξύ δηλαδή του το τέλους Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου. Έγιναν απόπειρε να πάνε κάποιοι να ζητήσουν, να συναντήσουν κτλ. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να φαίνεται λίγο δύο μήνε, αλλά σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την υπόθεση μάλλον είναι επίγον. Ε, έχουν γίνει κάποια διαβήματα, δράσεις, ενέργειες, ώστε να προσπαθήσουμε να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Θέλει κανείς άλλος να παρέμβει. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Um, thank you, Chair. Um, we mission, Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν ισχύουν οι συνθήκες για, για εκλογές. Ε, ακόμα και γίνονται τεχνικές βελτιώσεις. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με, πολιτικό, με το πολιτικό χώρο. Ε, δεν νομίζουμε λοιπόν ότι είναι σκόπιμο να στείλουμε αποστολή παρατήρησης εκλογών. Όπως είπαμε, Υπάρχουν ε, πολλοί, πολλοί οργανισμοί και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εργάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αιθιοπία. Έχουμε ε, συνεργασία με την Επιτροπή ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα για, με τον διαμεσολαβητή. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο πρόγραμμα, να, μεγάλος δρόμος να διανυθεί μέχρι να δημοκρατιστεί η χώρα αυτή. Ε, ε, πάντως το πρόγραμμα UNDP προβλέπει ε, στήριξη για τις εκλογές. Θέλουμε να βελτιωθεί το εκλογικό περιβάλλον, η διαφάνεια και η συμμετοχή, να, να, να αυξηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην Αιθιοπία μέσω της ε, παιδείας και ούτω καθεξή. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πριν να σκεφτούμε συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και επαναλαμβάνω ότι η συζήτηση συνεχίζεται, πάντως για την ώρα δεν ε, πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα όσον αφορά τη δράση της Ένωσης σε σχέση με αυτές τις συλλήψεις, σε αυτές τις συνεδριάσεις δεν μπορούμε να πούμε αυτά που λέμε στις διμερείς με τις, αρχέ με τις αρχές της Αιθιοπίας. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω ότι πάντοτε με ειλικρινή τρόπο μιλάμε για τα θέματα αυτά και παίρνουμε και ειλικρινές απαντήσεις από τους εταίρους μας, αλλά πάντως ε, αναφέρουμε ε, τα θέματα αυτά και τα συζητάμε σε επίπεδο Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών και είναι το βασικό μας ζήτημα συζήτηση στους τελευταίους μήνες και φυσικά θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και για θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της ΆΙΚΑΤ στη Νότιο Σουδάν οι δηλώσεις μας περισσότερο έχουν στόχο να λέμε δημόσια αυτά που συνήθως λέμε δια της διπλωματικής οδού, αλλά να αυξήσουν και την, τις γνώσεις του ευρέως κοινού για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Αυτό είναι ένα τμήμα της ε, ε, διπλωματικής μας σε σχέσεις με τις χώρες αυτές και όπως είπατε είναι Βρετανός υπήκος ο εν λόγω και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και να ζητάμε ότι, και μάλλον ό,τι μας ζητήσουν θα το έχουν. Ευχαριστώ. Η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξής. Όταν οργανώσαμε την ε, σημερινή συνεδρίαση, στραφήκαμε στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και στην Βρετανική κυβέρνηση και λάβαμε αυτή τη δήλωση, αυτή την ανακοίνωση που σας δώσαμε. Έχουμε λάβει και ενημέρωση σε σχέση ε, με το, μέχρι που μπορεί να φτάσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Πιστεύω ότι ίσως επειδή ένα από τα καθήκοντα που θέλουμε να έχουμε όσα υποεπιτροπή είναι η παρακολούθηση, η συνέχεια που μπορούμε να δώσουμε σε αυτά που κάνουμε εδώ, καλό θα ήταν ίσως να ξανασυναντηθούμε και να ξανασυζητήσουμε την περίπτωση ε, της Αιθιοπίας, ας πούμε, σε δύο μήνες από τώρα, και ίσως μέσα σε δύο μήνες να έχουμε καταφέρει να ενημερωθούμε για το ποια συνέχεια δόθηκε στην περίπτωση αυτή και στις άλλες περιπτώσεις που ετέθησαν σήμερα επιτάπητος από τις ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι νομίζω ότι αυτό έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να μιλάμε σήμερα και μόνο σήμερα για την Αιθιοπία και για το τι γίνεται σε κάποιες, με κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις υποθέσεις, αλλά και η Κομισιόν είναι καλό να ασχοληθεί με την παρακολούθηση αυτών των υποθέσεων. Επομένως, και βέβαια θα το δω με το Διευρυμένο Προεδρείο, τη Επιτροπή, αλλά καταρχήν θα έλεγα ότι μέσα σε δύο μήνε θα μπορούσαμε να δώσουμε το νέο μα ραντεβού για να συζητήσουμε για την Αιθιοπία και για τι συγκεκριμένε αυτέ υποθέσει που συζητήσαμε σήμερα. Και βέβαια η πρεσβεία τη Αιθιοπίας που εκπροσωπείται εδώ, φυσικά και έχει τη δυνατότητα να λάβει το λόγο εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, και μου δίνετε την ε, ευκαιρία να απαντήσω στα όσα υπόθηκαν από τα μέλη της ε, Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Από το 1995 η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ε, υποστηρίζει και διασφαλίζει τα δικαιώματα και ελευθερίας στα οπτικά μέσα. Στην Αιθιοπία υπάρχουν εκατοντάδες μέσα ενημέρωσης στην ε, Αιθιοπία. Έχουμε ε, και μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν ε, έρευνες ε, και δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Η κυβέρνηση συνεργάζεται μαζί τους για να τους δώσει δικαιώμα, να τους διευκολύνει. Τώρα, οι συλλήψεις των bloggers δεν έχει καμία σχέση με την, το επάγγελμά τους, αλλά λόγω, ε, λόγω υποψιών, έγιναν λόγω υποψιών για άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Ε, δεν μπορεί κανείς να μειώσει να δε, ή να αυξήσει τον χώρο του διαδικτύου έχουμε συγκεκριμένες ε, διατάξεις τις οποίες οφείλουν όλοι να ε, τηρούν. Όποιος και αν προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο θα δικαστεί. Το ιδιωτικό πρόβλημα με τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης της Αιθιοπίας, της είναι οι, το αποτυχάνουν να έχουν τη στήριξη του κοινού. Δεν μπορούν την καρδιά και την ψυχή του κόσμου. Και αυτό δεν μπορεί να καταλογιστεί ως έλλειψη πολιτικού χώρου. Οι, τα μέλη, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων είναι και εκείνοι ε, υπόλογοι στο, στους κανόνες δικαίου. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με τους ε, ε, φυλακισμένους μας, με τους κρατούμενους και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει καμία εξαίρεση με βάση το Σύνταγμά μας. Όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Η κυβέρνηση τους συνέλαβε διότι έχει αξιόπιστες πληροφορίες και αποδείξεις ότι έχουν παραβιάσει το δίκαιο και ότι έχουν αναμειχθεί σε εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, για την ε, έκδοση του κυρίου Αντεγκάζου Τσέγκε. Είναι γενικός γραμματέας ενός παράνο μιας παράνομης οργάνωσης. Είναι Βρετανός υπήκος και εκπαιδεύει στρατιωτικές ομάδες στην Ερυθρέα με στόχο να ανατρέψει την συνταγματικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Η οργάνωσή του έχει σαφώς ε, ε, ε, δηλώσει ότι θα διακόψει κάθε κυβερνητική δραστηριότητα εντός και εκτός της χώρας. Αυτό είναι έγκλημα ανώτατο επίπεδο. Όχι μόνο παραβιάζει το, το σύνταγμα της χώρας και πλήττει τη σταθερότητα της χώρας, αλλά είναι αδίκημα και υπό την Βρετανική δικαιοσύνη. Ενώ ταξίδευε για τις συνομωτικές του αυτές δραστηριότητα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σανά ε, και στάλει στην Αιθιοπία υπάρχει συνθήκη έκδοσης ανάμεσα στις δύο χώρες και εδώ δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Επί τη βάση της Σύμβασης της Βιέννης, μετά από αίτημα της Βρετανικής κυβέρνησης, του δόθηκε προξενική ε, πρόσβαση, μάλιστα εμφανίστηκε στην τηλεόραση και ήταν, ε, αντιμετωπίστηκε με πλήρη σεβασμό του δικαίου. Καταδικάστηκε από το ανώτατο δικαστήριο και τώρα η εκτέλεση της απόφασης εξαρτάται από τον επικεφαλής της χώρας. Για την ώρα κρατείται σε σοφρονιστήριο και γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματά του. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θέματα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την πολυμορφία μας και ο λαός μας αξίζει αυτή τη συμπεριφορά. Η δημοκρατία δεν μπορεί να ανθίσει μέσα σε αντιφάσεις. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της πρεσβείας. Θέλει κάποιος ε, το λόγο να ολοκληρώσουμε, θέλει κάποιος να πει κάτι. Όχι. Επομένως, το ραντεβού το ανανεώνουμε, παραλαμβάνω, για να ε, δούμε τι συνέχεια έχει δοθεί σε αυτή την υπόθεση και σε άλλες σχετικές. Σε δύο μήνες σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Vamos a pasar al siguiente punto de nuestro orden del día, que es el... Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξης, δηλαδή ανταλλαγή απόψεων για τον σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπαχρέν με τον Αμπίλ Ρετζάμπα, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τη Διεθνού Ομοσπονδία των Κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να να καλωσορίσω τέσσερι ε, ακτιβίστρε, ακτιβιστέ μάλλον από το Μπαχρέιν, που θέλω να τους καλωσορίσω. Είναι πίσω στην ναι, αίθουσα, στο βάθος. Ε, για να μην σα καθυστερήσω, σα δίνω μέσα στο λόγο. Thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ σε όλους για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και που βλέπω φίλους, βλέπω ανθρώπους που έχουν ε, κάνει δήλωση, τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες για την βελτίωση της κατάστασης στο Μπαχρέιν που ε, ε, ε, εγώ εκ μέρους του λαού μπορώ να σας πω ότι το εκτιμούμε ιδιαίτερος και το γεγονός ότι είμαι εδώ είναι επίσης ένας λόγος για τον οποίο σας σέβομαι γιατί ο ίδιος λόγος που με έφερε εδώ είναι και ο λόγος για τον οποίο ε, βρέθηκα στη φυλακή για δύο χρόνια για το γεγονός ότι άσκησα τα ανθρώπινα δικαιώματά μου ζητώντας την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων ή για, το, για τη συγγραφή απλών tweets. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Άννα Γκομές που με επισκέφτηκε στη φυλακή μαζί με άλλους ε, βουλευτές. Ευχαριστώ και τη Μέρι Σεκέλ, δεν ξέρω αν είναι εδώ, που θέτει το ζήτημα του Μπαχρέιν που το έχει θέσει το ζήτημα του Μπαχρέιν πολλές φορές και πολλές φορές ε, έχουν κάνει δηλώσεις για τον Μπαχρέιν σε διάφορες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από, αυτές τις, ε, ε, από αυτά τα ψηφίσματα για τον κόλπο. Όλες οι χώρες του κόλπου έχουν κυβερνήσεις που θεωρούν ότι μπορούν να αποφύγουν την κριτική λόγω της των οικονομικών σχέσεων που έχουν. Και εγώ βρίσκομαι εδώ για να σας ευχαριστήσω όλους και να πω ότι οι χώρες του κόλπου, ιδιαίτερα το Μπαχρέιν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το να είναι κανείς πλούσια χώρα, το να έχει κανείς οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σας ευχαριστούμε εσάς που εκθέσατε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν. Εγώ προσωπικά προ... κατάγομαι από χώρα όπου ε, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι. Ε, μια χώρα που δεν επιτρέπει την είσοδο ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν επιτρέπει την είσοδο ε, ομάδων ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και ευρωβουλευτών, για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως όχι κάθε φορά, αλλά τα ψηφίσματά σας και οι δηλώσεις που κάνετε ε, οδηγούν πολλές φορές και σε απελευθέρωση ανθρώπων. Στη δική μου περίπτωση, πιο σημαντική από την απελευθέρωσή μου ήταν το γεγονός ότι ήξερα ότι υπάρχουν άνθρωποι στο Ευρωκοινοβούλιο που, που με υποστηρίζουν στον αγώνα μου για τη, για τη δημοκρατία και, την, ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά ε, ενισχύουν τους ανθρώπους που παλεύουν στον Παχρέν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατάγομαι από μια χώρα που έχει ένα από τα πιο ε, καταπιστικά καθεστώτα. Ε, μια χώρα που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σύλληψης ε, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων. Από τη χώρα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτικών κρατουμένων που 17% του πλαθισμού της έχει περάσει από τις φυλακές τα τελευταία τρία χρόνια για το γεγονός ότι αγωνίζεται για την ε, δημοκρατία. που θεωρείται ότι είναι εχθρός του ίντερνετ από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα. η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη στην κατάσταση που, ε, από, στη χώρα που, ε, από την οποία κατάγομαι. Έχουμε 4.000 πολιτικούς ε, κρατούμενους σε μια χώρα που έχει πληθυσμό μικρότερο του ενός εκατομμυρίου. Δυστυχώς ε, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν κανονικότατες σχέσεις και κανονικότατες οικονομικές σχέσεις με τον Μπαχρέιν. Και είμαι εδώ για να ζητήσω από τους ανθρώπους και να τους πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα, κριτήρια, ε, αξίες που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Τμήμα των πολιτικών και των κοινωνικών μας συστημάτων, τμήμα των ε, ευρωπαϊκών οργάνων, των κατευθυντηρίες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη θανατική καταδίκη, για τις γυναίκες, αλλά όλες αυτές οι κατευθυντηρίες γραμμές δεν γίνονται σεβαστές από ορισμένες χώρες κατά, την, ε, ε, κατά τις οικονομικές δραστηριότητες με τον Μπαχρέιν. Θέλω να σα εμπιστήσω την, κατάσταση, την προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέιν. Να παρακολουθείτε τις χώρες που έχουν κανονικές σχέσεις με τον Μπαχρέιν δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν σχέσεις με αυτά τα, καταπιστικά καθεστώτα. Και όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν λάβει υπόψη ότι το ότι τμήμα ε, του πολιτικού σας συστήματος είναι και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα έπρεπε να έχετε οικονομικές σχέσεις με χώρες που ε, που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 90% των ακτιβιστών στον Παχρέν βρίσκονται στη φυλακή. Εγώ ήμουν ε, δύο χρόνια στη φυλακή. Απελευθερώθηκα πριν από τρία, τρεις μήνες. Και ε, οφείλεται σε ανθρώπους εδώ μέσα το γεγονός ότι έχω βγει πλέον από τη φυλακή θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία. Θα κάνουμε τον αγώνα που κάνατε εσείς πριν από πολλά χρόνια. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας σε δύο επίπεδα. Πρώτον, για να κατακρίνουμε τις χώρες που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα και να τους δείξουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Ευρώπης δεν είναι ανοιχτές για να κάνετε οικονομικές δραστηριότητες όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. αν παραβιάζετε τα πρότυπα αυτού του κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Είμαι ανοιχτό αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για να την απαντήσω. Σα ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σα ε, συγχαρώ ε, για την ε, μάχη που δίνετε. Να σα ευχαριστήσω και να σα ευχαριστώ και για την παρουσία σα εδώ. Κάποιος θέλει το λόγο. η Σίγουρα κυρία Γκόμες. Ναι, για να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου τις ευχαριστίες και να καλωσορίσω τον ε, κύριο Γαζάμπ εδώ. Τον είχα δει και με τον κύριο Χάρντ, την κυρία είναι και τον κύριο Ακουάτζα και τον κύριο Σαρίφ τότε είχαμε επισκεφθεί. Είδαμε πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση, πόσο άνθρωποι πόσο ο κύριος Ρατσά που ουσιαστικά αγωνίζονται για τα βασικά θεμελιώδη τους δικαιώματα και ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα καθεστώς που δεν είχε καμία διάθεση να ξεκινήσει ένα γνήσιο διάλογο, διότι η υπέρμαχη ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο πληθυσμός ο μεγαλύτερος πληθυσμός, το μεγαλύτερο μας πληθυσμό του Μπαχρέιν. Πάντως λήξη τη σύγκρουση είναι δύσκολο να υπάρξει και ίσω και κλιμάκωση είναι πιο πιθανό από αποκλιμάκωση. Είχαμε συναντηθεί και με κάποιου Αμερικανού εκεί. Έχει ο πέμπτος στόλος βάση στο Μπαχρέιν Uh, Υπήρχε ανησυχία για το τι γινόταν και απεσταλμένος των ΗΠΑ ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε απελαθεί, όπως και εγώ βέβαια προηγουμένως, από τον Μπαχρέιν. Υπήρχε πάντως τότε ελπίδα για διάλογο. Και ο διάδοχος του θρόνου ο πρίγκιπας προσπάθησε κάπως ε, να κάνει μια προσπάθεια, αλλά οι σκληροπυρνικοί τον ανέκοψαν. Νομίζω τώρα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος ε, Αλκουάτζα, που έχει έρθει εδώ στην Επιτροπή μας, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε από τη φυλακή και κατά πάσα πιθανότητα αυτό συνέβη χάρη στην κινητοποίηση της ε, διεθνή κοινότητας, Ο πατέρας του έχει ξεκινήσει απεργία πείνα, είναι στη φυλακή ακόμη, η αδερφή του συχνά μπαίνει στη φυλακή. Υπάρχουν παιδιά στη φυλακή, υπάρχουν πολλά έγγραφα. Αν πάει κανείς και μιλήσει τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ μίλησα με γιατρούς που τους απέλυναν το νοσοκομείο γιατί είχαν περιθάλψει <clears throat> θύματα της κρατικής βίας. Υπήρχαν άνθρωποι που χάσανε και την υπηκότητά τους με τον πλέον παράνομο τρόπο, χάνοντας και τα δικαιώματά τους. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον Μπαχρέιν και εγώ και άλλοι από την Επιτροπή εξεπλάγημεν όταν μία μέρα μετά από τις διαδηλώσεις είδαμε τη δήλωση της ε, ΕΙΕΔ που μιλάει για συγκράτηση από τους διαδηλωτές, τους ειρηνικούς αυτούς ανθρώπους. Αυτοί πρέπει να συγκρατηθούν. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Αν οι ειρηνικοί διαδηλωτές ε, μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι με τους καταπιεστές και τους καταστολείς. Υπήρχαν και στρατεύματα από τη Σαουδική Αραβία που είχαν έρθει για να τους ε, καταστήλουν τις διαδηλώσεις. Λοιπόν, θέλουμε να υπάρξει διάλογο στον Παχρέιν ε, με όλους. Ότι μπορεί να γίνει τον επόμενο μήνα, ε, ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Φυσικά και είναι μέρος της λύσης, ειρηνικής λύσης για το Μπαχρέιν. Αλλά εκλογέ μπορούν να γίνουν μόνο εάν υπάρχει και μια διαδικασία εθνική συμφιλίωση που να δρομολογηθεί, η οποία δεν έχει σε καμία περίπτωση δρομολογηθεί αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ζητήσουμε. Και αυτό χρειάζεται δράση από όλου μα. Και όχι μόνο από εμά, την Επιτροπή μα, το Κοινοβούλιο, την ΕΕΔ, αλλά και από τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη που συνεχίζουν σαν να μην τρέχει τίποτα, και εμπόριο όπλων κτλ. Πρέπει να υπάρξει εμπάργο εξαγωγής όπλων ε, σε χώρες ε, όπως αυτή που έχει προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι σε πολεμή ε, κατάσταση. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, Άννα. Θα δώσω το λόγο σε συναδέλφους πρώτα και μετά σε εσάς το λόγο. Λόχ Μπίλερ, καταρχάς. Ευχαριστώ μια ερώτηση που αφορά αυτούς τους 13 ε, ε, συλληφθέντες για την ε, δραστηριότητά τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκε ο Αμπτζάλα Ακαβάγια ότι σταμάτησε σήμερα την απεργία πείνας. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άλλοι ε, απεργοί πείνας. Και ένα ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερική Δράσης. Στο Μπαχρέιν δεν υπάρχει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ριάντ είναι αρμόδια και για το Μπαχρέιν. Και ακούσαμε μόλις πόσο σημαντικό ήταν το ε, γεγονός ότι οι συνάδελφοι ε, επισκέφτηκαν φυλακές. Θα ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον να, να ακούσουμε αν η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ριάντι είναι σε θέση να επισκέπτεται τακτικά τους φυλακισμένους και να παρακολουθεί και τις διαδικασίες. Και φυσικά ε, ο ε, πρέσβης ε, Κούλαχ είναι πάντοτε πολύ γρήγορας, γρήγορος όταν μιλούμε για φυλακισμένους, για κρατούμενους στη Σαουδική Αραβία, αλλά εδώ μιλάμε για γειτονική χώρα. Ευχαριστώ κυρία Παγάθα Ορτουντούα. Ναι, πολύ σύντομα ευχαριστώ πρόεδρε να σας συγχαρώ για μια ακόμη φορά γιατί ε, φέρετε στην Επιτροπή μας τόσο κατάφορες παρεμβάσεις των δικαιωμάτων για να μάθουμε και για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε ε, τον περιγυρό μας και με την Αιθιοπία αλλά και εδώ ε, το πρόβλημα είναι η στρατηγική που ακολουθούμε και επίσης υπάρχει και ε, σύγκρουση συμφερόντων. Ε, βλέπουμε και την δράση του Μπαχρέιν και της Αιθιοπίας των κυβερνήσεων. Πρέπει να συγχαρούμε το φιλοξενούμενο για το στένος του, την ανδρεία του, την αξιοπρέπειά του που συνεχίζει ε, να δραστηριοποιείται στον αγώνα του παρά τη δίωξη που, στην οποία υποβάλλεται εκεί που υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων, είτε από το κράτος είτε όχι, όποιος ε, αγωνίζεται ενάντια σε αυτές τις παραβιάσεις ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο αγώνας που δίνει είναι τεράστιος, χρονοβόρος, ε, με πολλά ε, εμπόδια. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία γιατί μόνο μέσα από την διεθνή κοινότητα ή από επιτροπές όπως η δική μας που υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να προέρθει κάποια βοήθεια, αλλά κυρίως η ισχύ των ακτιβιστών, η δική σας ισχύ είναι αυτή η οποία θα σας οδηγήσει μπροστά τα εμπρός. Είναι πολύπλοκος άγωνας που δίνεται και είναι σαφές ότι θα χρειαστούν χρόνια ε, για να επιτύχετε και δεν είναι και εγγυημένο ότι θα επιτύχετε. Το μόνο όμως που είναι εγγυημένο είναι ότι χωρίς μάχη δεν υπάρχει νίκη. Χωρίς αγώνα δεν υπάρχει το ενδεχόμενο της νίκης. Μας δίνεται ε, παράδειγμα με τη στάση σας. Ελπίζω να έχετε την εσωτερική δύναμη να συνεχίσετε. Και η διεθνής κοινότητα σιγά σιγά να μπορέσει να ασκήσει και αυτή η επιρροή για να αλλάξει το καθεστώς. Να βοηθήσετε εσείς που το κάνετε, αλλά να βοηθήσει και η διεθνή κοινότητα. Και να πάψουν αυτοί οι τοξικοί δεσμοί που υπάρχουν και να πάψουν να υποφέρουν οι λαοί. Βλέπω ότι έχουμε βέβαια όρια, περιορισμούς, γιατί αυτή η στρατηγική που έχουμε δεν μας βοηθήσει τόσο πολύ. Πάντως σας ε, ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Señora Pagaza Ortundúa, eh, Να δώσω τώρα το λόγο στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και μετά ο προσκεκλημένος θα ξαναλάβει το λόγο. Ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, είστε παρακαλώ. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για το αξίωμα που αναλάβατε. Είναι πολύ δύσκολα και ενδιαφέρον το αξίωμα που αναλάβετε και αν με επιτρέπετε θα περάσω στα αγγλικά για να σας πω αυτής εξ αρχής ε, ότι χαίρομαι πολύ που καλωσορίζουμε τον Αμπίλ Ρατζάντ εδώ ε, στο Κοινοβούλιο που τον βλέπουμε μεταξύ μας. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για όλους όσους έχουν συλληφθεί και κρατούνται για την ειρηνική συμμετοχή τους τις ειρηνικές τους δραστηριότητες στο Μπαχρέιν. Το κάναμε με δηλώσεις σε υψηλό επίπεδο και από την ίδια την είπατε εκπρόσωπο. Πριν έρθω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, και αν θέλουμε να καταλάβουμε καλά την κατάσταση στο Μπαχρέιν θα πρέπει να τη βάλουμε σε ένα πλαίσιο, σε ένα πολιτικό πλαίσιο και ιδίως στο σημερινό πλαίσιο ε, μετά τη ε, τις ε, συλλήψεις αυτές που έγιναν. Εγώ νομίζω ότι τα τελευταία γεγονότα δίνουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε όσους ε, ζητούν μια συμβαστική λύση που θα φέρει ένα, θα, θέσει ένα τέρμα σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Ο διάδοχος, ο πρίγκιπας, ε, έχει κάνει μια ανακοίνωση και εκεί αναφέρει τους τομείς μεταρρύθμισης θα μπορούσαν να μεταφερθούν ε, από την Εθνοσυνέλευση μετά τις εκλογές σε νομοθεσία. Ίσως να μην είναι τέλεια λύση, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί απόλυτα, πλήρως και αυτή είναι η έκκληση που απευθύνουμε σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να δράξουν την ευκαιρία δηλαδή, ώστε να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος ε, με καλή πίστη. Ο μόνος δρόμος για τον Παχρέν είναι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να συμμετέχει ε, η κοινωνία. Και πρέπει να το κατανοήσει αυτό και η κοινωνία στον Παχρέν και η διεθνής κοινότητα. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα βίας ε, τελευταία με τους αυτοσχέδιους εκριτικούς μηχανισμούς κυρίως και δράτω με της ευκαιρίας για να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει και θα συνεχίσει να καταδικάζει οποιαδήποτε χρήση βίας από οποιαδήποτε πολιτική δύναμη που τη χρησιμοποιεί ως μέσο πολιτικού διαλόγου. Ποτέ δεν μπορείτε να στηρίξουμε μια τέτοια πολιτική δύναμη. Και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι πιστεύουμε και πάνω από περισσότερο από ποτέ ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν ε, οι θεμητότατες αυτές τις ανησυχίες του Μπαχρέιν είναι η διεξαγωγή ενός ε, διαλόγου με πνεύμα συμφιλίωσης και θα πρέπει να αφαιθεί κατά μέρος ε, ε, ο σκληροπυρηνικός λόγος. Η πόλωση στον Μπαχρέιν, στην κοινωνία του Μπαχρέιν είναι, είναι ανυπόφορη και πρέπει να πάψει. Έχουμε τις συστάσεις του Μπίκη και υπήρξαν και κάποιες πρωτοβουλίε που ελήφθησαν για τη δημιουργία θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν ένα πρώτο βήμα. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι θεσμοί αυτοί θα πρέπει να δείξουν πλέον αυτά αποτελέσματα. Να δώσουν καλό παράδειγμα, να δημιουργήσουν τις απαραίτητες δομές για να φροντίσουν για την εφημερία του λαού του Μπαχρέιν. Ένα από τα θέματα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της ατιμορρησίας. Οι καταχρήσεις παρεμβάσεων των δικαιωμάτων, ε, οι θήτε πρέπει να προσαχθούν ενώπιν τη δικαιοσύνη. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είμαστε κατηγορηματικοί, είμαστε κάθετοι. Και ακόμα πιο ενδιαφέρον και πιο σημαντικό είναι σε αυτή την πολλωμένη κατάσταση που επικρατεί. Εμείς τι ζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε μια δέσμη μέτρων ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Και το πιο εύκολο που ζητάμε από την κυβέρνηση να πράξει είναι να εφαρμόσει πλήρω τις εστάσει UPR που τις δέχτηκαν. Να σα αναφέρω ορισμένου τομεί ανησυχία για εμάς. Ποινική δικαιοσύνη, παραδείγματο αποτροπή βασανιστήριων, προσαγωγέ, δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση, του συνεταιρίζεσαι, του συνέρχεστε, τη ε, ε, υπηκότητα, ηθαγένεια. Αυτά είναι ορισμένα μόνο, πολύ σημαντικά. Υπάρχει και μια ανεξάρτητη ε, επιτροπή που έκανε τι συστάσει αυτές και το υπήρξε και μια άλλη ανακοίνωση το 2014 το Σεπτέμβριο νομίζω. Και όλα αυτά τα έγγραφα δείχνουν τι χρειάζεται να γίνει στο τομέα των δικαιωμάτων στον Παχρέν. Πάντω υπάρχει και μια ακόμη πρόκληση η οποία είναι να γίνουν συγκεκριμένα βήματα στην υλοποίηση αυτών των συστάσεων και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, χτίζοντας πάνω στα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί μέχρι τώρα. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη άμεσα. Ιδίω για αυτού του κρατούμενου, αυτού του ειρηνικού ακτιβιστέ που είναι στι φυλακέ. Θα ρίνουμε την αντιπολίτευση να πάρει και το πολιτικό ρίσκο. Να ξαναπάρει τη θέση τη στο πολιτικό προσκήνιο και στου θεσμού. Να συμμετάσχει στι εκλογέ του Μάιο. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλιώς δεν πρόκειται να σπάσει αυτός ο φαύλο κύκλος. Επίσης, μια βιώσιμη συμβαστική λύση θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πιο θετικοί, συνθήκε συνθήκες για ε, τον εκδημοκρατισμό. Υπάρχουν ανοίγματα. Υπάρχουν συνταγματικέ μεταρρυθμίσει του 12. Υπάρχουν και προτάσει ε, που έκανε τώρα ο πρίγκιπας Όλα αυτά βέβαια πρέπει να τεθούν επιτάπητος, αλλά πρέπει πραγματικά ε, ο διάλογος να πάρει σάρκα και οστά και να μην επικρατήσουν οι σκληροπυρηνικοί. Πριν ολοκληρώσω, να σας πω, απαντώντας ε, στην κυρία Λόχ Μπίλερ, εμείς δεν έχουμε πράγματι αντιπροσωπεία στο Μπαχρέιν. Αυτό είναι μειονέκτημα Έχουμε όμω μια αντιπροσωπεία στο Ριάτ και προσπαθούμε να καλύψουμε και τον Μπαχρέν. Και ο πρέσβη και όλοι οι συνάδελφοι τη αντιπροσωπεία εκεί προσέχουν πάρα πολύ την κατάσταση στον Μπαχρέν, επισκέπτονται τη χώρα πολύ συχνά. Και άλλοι υπάλληλοι και ο ειδικό εκπρόσωπο μετέβη στον Μπαχρέν, μίλησαν ανοιχτά. Ζήτησε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στον κόλπο, όπω ξέρετε. αρχίσαμε με ενθαρρύνουμε διπλωμάτες να παρακολουθούν, ε, να είναι παρατηρητές σε δίκες. Είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στον τομέα αυτό. Και τώρα ολοκληρώνω, κύριε Μπρό, και λυπούμε που καταχράστηκα του χρόνου σας και στον κύριο ε, Φωμέ λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε λύση η οποία θα ε, υπαγορεύεται από τους κατοίκους του Μπαχρέν και θα έχει στόχο την εφημερία του λαού του Μπαχρέιν. Presses ahead for key reforms and the need for reconciliation. Thank you so much for your time. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αλεξανδρίδης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεξανδρίδη. Θέλετε να κάνετε τώρα ερώτηση, κυρία Γκόμες. Το φίλο μας, τον εκπρόσωπο της ΕΕΔ, Θέλω να τον ρωτήσω. Αυτή η δήλωση της Λέδης Άστον που ζητά την απελευθέρωση των κρατουμένων, από πότε χρονολογείται, γιατί εγώ δεν έχω δει καμία. Κάποιες δηλώσεις που ζητούν εθνική συμφιλίωση, να παίξουν πολιτική διαδικασία κτλ. Έχω δει. Αλλά συγκεκριμένα να ζητείτε απελευθέρωση των κρατουμένων δεν έχω δει. Ή τώρα ή πιο μετά έχετε την καλοσύνη να με ενημερώσετε. Κύριε Αλεξανδρίδη, λέει πρόεδρος. Αναφέρομαι στην δήλωση της κυρίας Άστον της 16ης Αυγούστου 2012, ευκαιρία, μάλλον με την, ε, στην περίπτωση της καταδείξης του κυρίου Νατσάπ. Δεν μίλησα όμως μόνο για αυτόν, αλλά για όλους τους πολιτικούς κρατουμένους. Όλους τους κρατουμένους συνείδησης. Υπήρξαν και ιδιωτικές ε, προφορικές δηλώσεις κυρίας Άστον πέρυσι, μετά από την υπουργική GCC που έγινε στον Παχρέν και εκεί μίλησε και πάλι για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ήταν καλά προετοιμασμένος ο κύριος Αλεξανδρίδης, ε? λέει η πρόεδρος. Αν συμφωνείτε, θα δώσουμε το λόγο σε έναν από τους ακτιβιστές που ήρθε από τον Παχρέιν. Πέντε λεπτά μόνο έχουμε δυστυχώς τη διάθεσή μας, αλλά θα θέλαμε έστω κάποιον από αυτούς να ακούσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χουστέιν Αμπτούλα, είμαι ο εκπρόσωπος του Americans for Democracy στο Μπαχρέιν. Σε πέντε λεπτά θα προσπαθήσω να καλύψω τα ζητήματα που έχουν ε, τεθεί εδώ από τους ομιλητές. Είναι πολύ σημαντικό για μας το γεγονός ότι μας προσκαλέσατε εδώ σε αυτήν την ε, υποεπιτροπή για να εκφράσουμε και εμείς τη δική μας ε, γνώμη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στη χώρα μας, στο Μπαχρέιν όπου αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα ε, η δική μου ηθαγένεια ε, ανακλήθηκε για τις εκλογές. Συμφωνώ απόλυτα με τον ε, κύριο της ε, Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρέπει να δράξουμε κάθε ευκαιρία και που προσφέρεται από την ε, κυβέρνηση του Μπαχρέιν για να επιληθεί η κατάσταση. Η κατάσταση αυτή που υπάρχει εδώ και 3,5 χρόνια και οδεύουμε προς τον τέταρτο χρόνο πλέον. Αν πράγματι είναι μία λύση και όταν σπούδαζα και ε, σπούδαζα για την ιστορία των χωρών της Ευρώπης, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, οι εκλογές δεν είναι πάντοτε, δεν είναι η λύση, είναι το αποτέλεσμα λύσεων. Αυτό που χρειάζεται τον Προχρέιν αυτή τη στιγμή είναι μια άμεση διαδικασία συμφιλίωσης και οικοδόμηση μέτρων ε, εμπιστοσύνης, ε, απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Δεν μπορούν να γίνουν επιτυχημένες εκλογές όταν η μισή αντιπολότευση που ξεκίνησε το, το, το κίνημα, την επανάσταση του, της 14ης Φεβρουαρίου ε, δεν μπορείς να έχεις επιτυχημένες εκλογές όταν υπάρχει, ε, όταν υπάρχει διέρεση της χώρας στη βάση ε, θρησκευτικών διαιρέσεων, δεν μπορείς να έχεις επιτυχημένες εκλογές όταν υπάρχουν βασανιστήρια στη χώρα. Όταν πολιτικοί κρατούμενοι αυξάνονται. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διάλογος, σοβαρός διάλογος χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεση για να μην ξανάρθουμε μετά από πέντε χρόνια για να ξανασυζητήσουμε τα ίδια ζητήματα ότι το Μπαχρέιν δηλαδή έχει πολιτικά προβλήματα. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν διαρκώς όταν συζητούμε για το Μπαχρέιν. Φυσικά κατανοούμε πλήρως και χαιρετίζουμε κάθε θετικό βήμα που θα αναλάβει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν ε, έτσι χαιρετήσαμε το, τη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος του Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες κινήσεις. Αυτό που κάναμε ήταν... Ε, το HRB είναι η δική μου μη κυβερνητική οργάνωση και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και μάλιστα εκθέσαμε μια, ε, δημοσιεύσαμε μια έκθεση στην οποία υπάρχουν 30 ε, καταγγελίες προς τον συνήγορο του πολίτη και θέλαμε να δούμε αν τελικά διερευνήθηκαν οι υποθέσεις αυτές και διαπιστώσαμε ότι ακόμη κανένας δεν έχει επικοινωνήσει με αυτά τα θύματα. Οι υποθέσεις τους δεν έχουν διερευνηθεί. Η μόλι απάντηση που λάβαμε από τον συνήγορο του πολίτη ε, ήταν ε, να μας ρωτήσει ποιος ακριβώς είναι, ποια, ακριβώς είναι το, το σημείο επαφή σας ε, στη χώρα εμείς και για λόγους εμπιστευτικότητας δεν μπορούσαμε να δώσουμε τέτοια στοιχεία. Οπότε ξαναλέμε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι μακροπρόθεσμη ε, λύση. Επίσης, οι στάσεις UPR που μάλιστα έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν ε, βρίσκονται όλα σε μια έκθεση που έχω εδώ μαζί μου. Η κυβέρνηση του Μπαχρέιν μέχρι σήμερα δεν έχει... Ε, εφαρμόσει την πλειονότητα των ε, συστάσεων ε, αυτών. Σύμφωνα με το State Department, σύμφωνα με ε, διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι δικές μας εκθέσεις δεν έχουν υλοποιηθεί. Το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν λέει το ίδιο, έχει την ίδια άποψη. Και να τελειώσω λέγοντας ότι η κοινότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Παχραήν θα ήθελε πραγματικά πάρα πολύ να, βρει, να βρεθεί μια λύση στη χώρα. Έρχονται με ανοιχτά τα χέρια και ανοιχτά την καρδιά τους λέγοντας στην κυβέρνηση του Παχραήν ότι η καλύτερη λύση είναι μια λύση που θα ε, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και που θα περιλαμβάνει βεβαίω απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κανείς άλλος να καταφέρει να πει σε τόσο σύντομο χρόνο τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στο προσκεκλημένο μας και με το σημείο αυτό ολοκληρώνω και με την δική του παρέμβαση ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της μέρης της διάταξης. Θα μπορούσα να προσθέσω κάποια πράγματα, αλλά συγκεκριμένα ως προς την παρουσίασή σας που είναι ακριβώς η, η, ο τρόπος με τον οποίο η Βρετανική κυβέρνηση ε, ε, παρουσιάζει τα πράγματα στον κόσμο. Και Μόνο έτσι θα μπορούσαν άλλωστε να γίνουν τα, τα πράγματα. Με κάθε σεβασμό στην ε, Βρετανική κυβέρνηση και τη Βρετανική κοινωνία, όπου εμείς ε, μάθαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να πω ότι πολλές φορές ε, υπάρχει μια διαστρέβλωση όσον αφορά την κατάσταση του Μπαχρέιν. Εμείς θέλουμε πολιτική λύση, δεν θέλουμε να... Θέλουμε, δεν, θέλουμε, δεν ζητάμε εκλογές αγνώντας ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει διάλογος. Πρέπει, λοιπόν να σας ζητήσω να ζητήσετε από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να έρθει σε συνεννόηση και σε διάλογο με την αντιπολίτευση. Αυτό που έγινε τώρα είναι ότι το, ο, Βασίλης, ο βασιλιάς αποφάσισε ότι θα γίνουν εκλεγές. Θέλετε δεν θέλετε. Αυτός δεν είναι ο τρόπος. να αντιμετωπίζει κανείς ανθρώπους που εκπροσωπούν το 15-18% του πληθυσμού. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση θα πρέπει να καθίσουμε μαζί για να εξέλθουμε από αυτή την κρίση. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ και ευχαριστώ βεβαίως και την, ε, το, γραφείο της ΥΠΑ της εκπροσώπου που ζήτησε την ε, ε, απελευθέρωσή μου. Ξέρετε ότι ε, μιλούμε για τον Αμπτουλά ο οποίος είναι ε, υπήκος του Μπαχρέιν και υπήκος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος βασανίστηκε και μάλιστα χρειάστηκαν 16 βίδες για να συγκρατήσουν το πρόσωπό του και πλάκες από ατσάλι για τον ίδιο σκοπό και είναι ένας από τους χιλιάδες ε, κρατούμενους, φυλακισμένους αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις. Αυτό που λέμε με κάθε σεβασμό βεβαίως ε, είναι ε, ναι, απελευθερώστε τους ε, πολιτικούς κρατούμενους. Το 60% των ηγετών βρίσκονται στη φυλακή. Σταματήστε τις διακρίσεις, την περιθωριοποίηση, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. αυτών που εκπροσωπούν το 17% του πληθυσμού. 17% και η εκπροσώπησή τους στα, στα θεσμικά όργανα και στο στρατό είναι 0 και 1%. Πρέπει να υπάρχουν νόμοι. Η κυβέρνηση του, Μπαχρο, του Μπαχρέιν αρνείται. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν έχει ε, νόμο που να λέει ότι οι διακρίσεις είναι έγκλημα. Ακόμα και αν περάσει ένας τέτοιος νόμος από το Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση τον απορρίπτει. Δεν μπορείς να, όλες οι, οι εξουσίες να βρίσκονται στα χέρια ενός ανθρώπου, η δικαστική, η εκτελεστική, η νομοθετική εξουσία. Ένας άνθρωπος να αποφασίζει για τα πάντα. χθες ε, ελήφθη μια απόφαση να μειωθεί ο αριθμό των κυβερνητών, έτσι, χωρίς να ξέρει κανείς. Εμείς ως ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέμε ότι θέλουμε πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέλουμε κριτήρια για τον ίδιο σκοπό, θέλουμε κατευθυντήρε γραμμές, οι οποίες να τηρούνται. Πώς? Δεν μα νοιάζει. Ο Πρωθυπουργό, όπω γνωρίζετε, Ξέρετε ότι έχουμε τον ίδιο Πρωθυπουργό εδώ και 42 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην βασανίζονται άνθρωποι. Και πολλοί άνθρωποι μάλιστα βασανίστηκαν μέχρι θανάτου. Η βία φυσικά ε, πρέπει να γίνει, είναι καταδικαστέα από όλους μας. Αλλά θα πρέπει να πούμε ποιο είναι ο θήτης εδώ πέρα. Ε, το, το Μπαχρέιν, η κυβέρνηση του Μπαχρέιν έχει σκοτώσει 150 ανθρώπους με δακρυγόνα, με, με σφαίρες, με εξοπλισμό ε, καταστολής ε, διαδηλωτών που έχει εισαχθεί από την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν είναι η έκθεση. Αλλά τι αφορά αυτή η έκθεση. Αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, τους τελευταίους δύο μήνες. Δεν μιλάμε για την όλη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Μπαχρέν. Μιλάμε μόνο για αυτούς τους δύο μήνες. Και υπάρχει αυτό το θετικό αίτημα. Αλλά να σας πω κάτι. Το 17% των ανθρώπων που ε, δολοφονήθηκαν μετά την ε, δημοσίευση αυτής της έκθεσης εκείνη τη στιγμή υπήρχαν χίλιοι πολιτικοί κρατούμενοι. Και αντί τελικά να μειωθούν και να απελευθερωθούν μάλλον αυτοί οι πολιτικοί κρατούμενοι, σήμερα έχουμε 4.000 κρατούμενους. Άρα το ζήτημα δεν είναι να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει συνήγορος του πολίτη κτλ. Είναι να υπάρχει η πολιτική θέληση, διότι υπάρχουν θεσμικά όργανα αλλά δεν έχουν αρμοδιότητες εμείς όταν ε, βλέπουμε ανθρώπους μετράμε τι γίνεται κάτω στον κόσμο, όχι τα μεγάλα λόγια που ακούγονται. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ανοίξαμε γραφεία εδώ στις Βρυξέλλες για να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι εσείς είστε το, το θεσμικό όργανο με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο και θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή σε εσά για να σταματήσουν αυτοί να διαστρεβλώνουν την, ε, την κατάσταση και να, παρα, και να ενημερώνουν εσφαλμένα την, την κοινή γνώμη. Για, για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ε, ζητούμε τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε βεβαίως και για την υποστήριξη όλων των προηγούμενων ετών. Την εκτιμούμε απόλυτα και την χαιρετίζουμε. Και ε, ξέρω ότι χιλιάδες άνθρωποι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέω σήμερα εδώ είναι που με έφεραν στη φυλακή για δύο χρόνια και αυτό που σας ζητώ είναι να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Να, ε, να κάνουμε πράγματα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην, ε, στο Μπαχρέιν. Τα ανθρώπινα, πρέπει να τους πούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να γίνονται σεβαστά παντού. Και πρέπει να σταματήσουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει σκοπό να τα παραβιάζει. Και συγγνώμη που μακρηγόρησε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Ε, πρέπει να απουσιάσω αλλά έχουμε την Αντιπρόεδρο, την κυρία Λόχμπιλερ μαζί μας, η οποία θα πάρει τη σκητάλη μέχρι το τέλος της συνεδρίασης και θα συμπληρώσει κάτι στα διάφορα. Κυρία Λόχμπιλερ, το είχε πει το πρωί. Έχετε κανένα δύο σημεία να διεκπαιρεώσετε ακόμα λοιπόν και μετά θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Είδα το που δεν το ξέχασα κυρία Λόχμπιλερ. Από μένα καλό βράδυ.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 So, colleagues, then we continue. Ωραία συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το δίκτυο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, σχετικά με την ετήθησια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλώς ορίσατε όλοι, τόσο ως δίκτυο, αλλά όσο και ως μεμονωμένες οργανώσεις που συμβάλλεται στην κριτική που ασκείται, στα στοιχεία που συλλέγονται που και εμείς θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και να αξιοποιήσουμε στις εργασίες μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως κάθε χρόνο εδώ στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε ήδη λάβει την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο ε, την πρόσκληση της Κομισιόν για τη σύνταξη αυτής της ε, έκθεσης και ενημερωθήκαμε ε, ότι ο Αντώνιο Παντσιέρη θα είναι ο εισηγητής φέτος από τους σοσιαλιστές. Επίσης, έχουμε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναδιαρθρώθηκε με βάση το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης βρισκόμαστε επισήμως ή ανεπισήμως ε, στις πολιτικές ομάδες στην διαδικασία και στις ε, συζητήσεις με το EAS για το ποια θα είναι η μορφή της, ε, του νέου αυτού σχεδίου δράσης που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Οπότε θα σας ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Είναι μαζί μας η κυρία Ζακλίν Χολ, εκπρόσωπος ε, του δικτύου συνολικά. Έχουμε την κυρία Γκέλ, του Σεπούλκρε. Συγγνώμη, νο, ξέρω ότι από την προηγούμενη φορά έπρεπε να το είχα μάθει το όνομά σας είναι η Λότε Λάιχτ από τη Human Rights Watch εδώ στην, ε, στις Βρυξέλλες, Κατρίν Τεντέριαν από τη Διεθνή Αμνηστία και βλέπετε ότι δεν είναι ισορροπημένο προς, το φύλλο ε, το πάνελ μας, αλλά ε, παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε. Ε, θα ήταν επίσης καλό να σας ακούσουμε εσάς πρώτα και στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ο, για, την, για να ξεκινήσει η συζήτηση ο κύριος Αντώνιο Παντσέρη. Κυρία Χολ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Τρόικα του Δικτύου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που όπως γνωρίζετε είναι ένα δίκτυο που συμπεριλαμβάνει 48 ε, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε όλη την Ευρώπη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε εδώ. Ε, οι συνάδελφοί μας, οι υπερασπιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα μας έχουν πει επανειλημμένως για το πόσο εκτιμούν την δράση του Κοινοβουλίου για την ε, υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το γεγονός ότι μπορεί πραγματικά το Κοινοβούλιο και οι απόψεις που υιοθετεί να σημάνει τη ζωή το θάνατο για πολλούς ανθρώπους, πολλούς κρατουμένους. Σας ευχαριστούμε. Επίσης, ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σχέση μας με αυτήν την ε, Επιτροπή για το γεγονός ότι ε, καλή σε λογοδοσία τις άλλες ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ε, για παράδειγμα η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που ετοιμάζει την στρατηγική της αυτό το φθινόπωρο. Και ανυπονομονούμε να δούμε βεβαίως και την ετήσια έκθεση, την φετινή. Από αυτή την άποψη προσβλέπουμε και σε αυτήν την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο εντός του Κοινοβουλίου για την υπεράσπιση των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δει τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραβιάζονται ή να ε, δέχονται επίθεση ακόμη και εδώ μέσα και θέλουμε η Επιτροπή αυτή να είναι στην καρδιά του αγώνα ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραμείνουν στην καρδιά της ε, Ευρώπης Οπότε θέλω να αναφερθώ σε τέσσερις τομείς δράσης σας, όπου βλέπουμε ότι στο, στο δίκτυό μας ότι μπορούμε να σας υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε όσους υπέγραψαν την έκκλησή μας για ε, τις ευρωεκλογές για τα ανθρώπινα δικαιώματα Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανάγκη να ε, γίνει κύριο ζήτημα ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στο Κοινοβούλιο. Πώς θα το κάνουμε αυτό, να ε, λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόψη του τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συζητούνται το θέμα αυτό όχι μόνο εδώ σε αυτή την Επιτροπή αλλά και σε άλλες επιτροπές όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η Επιτροπή Ανάπτυξης. Επιτροπές οι εργασίες των οποίων σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα θέλαμε κάθε επιτροπή και κάθε αντιπροσωπεία να έχει τουλάχιστον ανεπισήμως έναν αντιπρόεδρο με αρμοδιότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Και θέλουμε τα, μέλη αυτής της Επιτροπής να ασκήσουν πιέσεις στους συναδέλφους στις πολιτικές ομάδες για αυτόν τον σκοπό. Δεύτερον, θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να επιδιώξει μια ε, συνεργασία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία με τα εθνικά κοινοβούλια. Να γίνονται τακτικές ε, συνεδριάσεις, να ε, συζητώνται επίγοντα ζητήματα και να αναλαμβάνονται δράσεις ώστε να υπάρχει συνεκτικότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Τρίτον, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι ότι αυτή η Επιτροπή μπορεί να ε, αποκτήσει επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Είναι και η οι τοποθετήσει που ακούσαμε, αλλά αφορά αυτό που λέω και τις ε, επισκέψεις σε τρίτες χώρες πάντοτε να γίνονται συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών και με ανεξάρτητες οργανώσεις. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων ε, στις τρίτες χώρες. Επίσης, να διασφαλίσουμε ότι τα ψηφίσματα ε, πήγοντος χαρακτήρα θα πρέπει να, να, να παρακολουθούνται και να πω ότι η διατύπωση ε, σε αυτά τα ψηφίσματα θα πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα, μηχανισμούς παρακολούθησης, ανθρώπους που θα ε, συνεχίσουν την, ε, την παρακολούθηση της, της εκάστοτε κατάστασης. Και τέλος, θεωρούμε ότι η Επιτροπή αυτή παίζει σημαντικό ρόλο στην ευθυγράμμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής με το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Σκεφτόμαστε, έχουμε στο νου μας και τις κυρώσεις σε τρίτες χώρες Συνόδου ε, συνόδους κορυφής ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε, χώρε όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Σα ευχαριστούμε και πάλι που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ. Η Επιτροπή σα είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την διαφάνεια και τη λογοδοσία για το πώ υλοποιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Είμαστε μαζί σας, θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουμε ώστε ε, το ευρωπαϊκό όραμα να διατηρήσει στην καρδιά του τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο στην Γκίλ. Uh, Thank you. So uh, I would to uh, σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω καταρχήν στην πραγματικά, πραγματική προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για τα Ανθρώπινα και τη Δικαιώματα και τη Δημοκρατία που υιοθετήθηκε το 2012 από την Ένωση και το πώς μπορεί πραγματικά να εξυπηρετήσει την βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τόπου και στις διάφορες ε, ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορεί επίσης να ε, βελτιώσει την ποιότητα της αναφοράς, που, των εκθέσεων μάλλον που κάνει η ίδια η Ένωση για τις δραστηριότητες της. Με αυτό ως σημείο εκκίνησης θα ήθελα να τονίσω Κάποια σημεία τα οποία αναπτύχθηκαν στην έκθεση του Συμβουλίου του 2013 για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να επιμείνω για το γεγονός ότι αν είχαμε πραγματική πρόοδο θα πρέπει να υπάρξει και βελτίωση στην πράξη και στις ε, ε, αναφορές, στις σχετικές εκθέσεις που συντάσσει η κυρία Άστον και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε πραγματικά να αντιμετωπιστούν τα βασικά προβλήματα που παραμένουν, που επιμένουν στο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για κάποιες γενικές δεσμεύσεις της Ένωσης. Καταρχήν, ε, αν μιλήσουμε για την αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά και κάποια θέματα όπως ε, μετανάστευση και αντιτρομοκρατική δράση. Για τις αξιολογήσεις ε, αντικτύπου έγιναν κάποιες απόπειρες από την Ένωση να εισαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις αξιολογήσεις τέτοιου τύπου πριν να γίνονται σημαντικές πολιτικές ή δραστηριότητες. Στην έκθεση του Συμβουλίου του 2014 τονίζεται ότι αυτό έχει επιτευχθεί, αλλά εμείς δεν συμμεριζόμαστε αυτήν την αξιολόγηση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου δεν έχει γίνει επαρκής ε, αξιολόγηση του αντικτύπου ούτε έχει γίνει από ανεξάρτητο συνεργάτη. Ε, η προστασία των επενδύσεων, για παράδειγμα, ποτέ δεν έχει εξελογηθεί και είναι πραγματικά πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα λόγω του αντίκτυπου που μπορεί να έχει όχι μόνο στις ξένες χώρες αλλά και στην Ένωση. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη Ε, της ε, και την της επιμονής μας ε, στην ποιότητα αυτών των, μελετών αντικτύπου. Είδαμε, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις για την Κίνα ή για τη Βυρμανία, όπου η Κομισιόν λέει ότι επειδή πολλαπλασιάζει τους επενδυτές, τα δικαιώματα, μάλλον τα ιδιοκτησιακά των επενδυτών, που συμβάλλει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση και πρέπει να διορθωθεί. Σε σχέση με τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, η έκθεση για την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 2013 ε, τονίζουμε μόνο ότι δεν αρκεί και θα ήθελα να καταγράψουμε την, τη μελέτη του Λοράν Μπαρτέλ που λέει ότι <coughs> οι ρήτρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πλήρως ανεπαρκείς για να αντιμετωπιστούν ε, τα, σωστά, τα, τα, τα σοβαρά αυτά θέματα. Τώρα, λίγα λόγια Όσον αφορά το στρατηγικό πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό στις μελλοντικέ εκθέσεις του Συμβουλίου και της Άστον και το διαδοχό τη και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση και καλύτερη περιγραφή των όσων ε, γίνονται συγκεκριμένα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών. Έχουμε δει πολλές δραστηριότητες ε, ας πούμε στο πλαίσιο της μετανάστευσης ή στην ε, ε, αντιτρομοκρατική δράση που έχουν σημαντικό αντίκτυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω τώρα το χρόνο για να τα πω όλα, να πω σε όλες τις λεπτομέρειες, γι' αυτό θα σταματήσω σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε το Human Rights Watch σε αυτή τη συνεδρία. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εμείς συμφωνούμε απόλυτα ε, με το HRDN. Είμαστε και περήφανα μέλη του δικτύου αυτού. Συμφωνούμε με όλα όσα είπε η Ζακλίν Πιστεύω ότι μπορεί το Κοινοβούλιο να τα εφαρμόσει όλα αυτά εύκολα και να κάνει έτσι πραγματικά τη διαφορά. Σας παρακαλώ λοιπόν να λάβετε πολύ σοβαρά αυτές τις συστάσεις και να τις υλοποιήσετε. Θα ήθελα τώρα τα λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου ε, να τα αφιερώσω στο να σας ε, κάνω ε, μία έκκληση να ζητήσετε την απελευθέρωση των υπεμάχων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, κρατωμένων συνείδησης. Ε, πρέπει να γίνει ένας μεγάλος στόχος σας η απελευθέρωσή τους. Ε, ακούσατε έναν από αυτούς και στον Παχρέιν τον έβαλαν φυλακή γιατί αυτά που λέει δεν τους αρέσουν και προκαλεί το μονοπόλιο που έχουν στην εξουσία και την ατιμορρησία με την οποία κυβερνούν και ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τους ίδιους τους, τους συμπολίτες. Αναφέρθηκε το στρατηγικό πλαίσιο, εγκρέθηκε τον Ιούνιο 25 Ιουνίου του 2012 και θεωρούμε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό εργαλείο μια υπόσχεση που δίνει η κυβέρνη, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για όσους ε, ειρηνικά αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το στρατηγικό πλαίσιο συγκεκριμένα λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει πλήρω αυτού που συνηγορούν υπέρ τη ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία και των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι ο ρόλο του Κοινοβουλίου δύο χρόνια μετά και τη Επιτροπή σα είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να τηρούν την υπόσχεση αυτή, τη δέσμευση αυτή και οι υπάλληλοι να λογοδοτούν για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν ε, ή δεν εφαρμόζουν την υπόσχεση αυτή, τη δέσμευση αυτή, ιδίω σε σχέση με τους ε, ακτιβιστές που κρατούνται στις φυλακές όλο τον κόσμο. Χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ε, μια ανακοίνωση, χειρή ανακοίνωση, μετά την απόφαση Κινέζικου Δικαστηρίου για... Ε, να φυλακίσει η φόρου ζωή στον νόημα ότι έναν Ουιγούρο, Κινέζο, ακαδημαϊκό, που τι έγκλημα διέπραξε. Ήταν υπέρ του διαλόγου μεταξύ των ε, διαφόρων κοινοτήτων. Και αυτό ερμηνεύτηκε από το Κινέζικο Δικαστήριο ως αποσχιστικό ε, και γι' αυτό τον έβαλαν φυλακή για όλη του τη ζωή. Ε, ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταδίκη αυτής της απόφασης, την οποία θεώρησε αδικαιολόγητη εντελώ και απαιτεί την άμεση ανεφόρον απελευθέρωση. Το ανθρώπου αυτού, Human Rights Watch, ε, χαιρετίζει τέτοιες εκφράσεις αρχών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζει να γίνουν και τα επόμενα βήματα ώστε το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη και τα κράτη-μέλη της Ένωσης να ενώσουν τις δυνάμεις τους ε, για να ασκήσουν ε, πιέσεις στην Κίνα ώστε να απελευθερώσει τον ε, τότη. Και τώρα, και εδώ είναι η δυσάρεστη είδηση, αυτή η χειρή ανακοίνωση που είδαμε χθε δεν είναι αντίστοιχη σε αυτά που συνήθως βλέπουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ένας θαραλέος, ακαδημαϊκός, ακτιβιστής, προσπιστής των ανθρώπινων δικαιωμάτων μπαίνει φυλακή. Πράγματι, είναι σπανιότατο το φαινόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητεί απελευθέρωση κάποιου, τέτοιου κρατουμένου και συνεχώς με αποφασιστικότητα να επιδιώκει αυτό το, την απελευθέρωση και τα αποτελέσματα μιλούν και από μόνα τους κατά κάποιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έβγαλε κανέναν από τη φυλακή ουσιαστικά. Πρόσφατα μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζήτησε την απελευθέρωση του πλέον γνωστού ακτιβιστή του Μπουρούντι του Πιέρ Κλαβιέρ που ε, δικάζεται. Ούτε την απελευθέρωση του Λέλα, της Λέλα Γιάννους από το Αζερμπαϊτζάν που πολλοί από εσάς ε, ε, έχετε ψηφίσει να είναι υποψήφιοι για το βραβείο Ζαχάροφ. Ούτε παρά τα όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σαφής στις εκκλήσεις της για την ανεφόρον άμεση ε, απελευθέρωση του Αμπτούλ Χαντί Αλκαβάτσα και άλλων στο Μπαχρέιν. Άρα, το να βγουν από τη φυλακή οι πολιτικοί κρατούμενοι δεν φαίνεται να ήταν προτεραιότητα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Αν κρίνουμε απλά και μόνο από τις δηλώσεις και όμως και από τις συναντήσεις που είχαμε με διπλωμάτες που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να έχει μια στρατηγική για να επιδιώξει την απελευθέρωση ακτιβιστών. Ούτε και τη θέσμευση φαίνεται να έχει γι' αυτό. Ούτε και είχε και μεγάλη επιτυχία στις προσπάθειες να βγάλει ακτιβιστές από την ε, φυλακή. Εγώ σας, βοηθώ, σας ζητώ να βοηθήσετε να αλλάξει αυτό. Να γίνει μια νέα αρχή τώρα. Έχουμε ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια νέα Επιτροπή Ευρωπαϊκή, νέο Πρόεδρο του Συμβουλίου και μια νέα επατή εκπρόσωπο. Έχουμε λοιπόν μια νέα ευκαιρία στους κρατούμενους επασπίσεις των δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο να τους δείξουμε ότι κάτι σημαίνουν και ότι η προθυμία τους, η ετοιμότητά τους να ε, αγωνιστούν για τη δημοκρατία είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει και εμείς να κινήσουμε γη και ουρανό για να τους βοηθήσουμε. Σας ε, ευθύνω έκκληση λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνετε την απελευθέρωση αυτών των κρατουμένων βασική προτεραιότητα, βασική μέρημνα και να ξεκινήσετε και στις ακροάσεις τώρα που θα έχετε, ξεκαθαρίζοντας αυτό και στους νέους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην νέα ΥΠΑΤΗΚ πρόσωπο. Και σας παρακαλώ να τους ρωτήσετε να σας απαντήσουν πώς θα συνεργαστούν μαζί σας ε, για να τιμήσουν ε, αυτή την δέσμευση που ανέλαβε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μόνο του, το είπε η Ζακλίν, ίσως έχω μακρηγορήσει για πολύ, αλλά μου δίνετε ένα ακόμη λεπτό. Μπορεί λοιπόν και έχει και κατά τον παρελθόν βοηθήσει σημαντικά αυξάνοντας ε, την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης, έδωσε ονόματα, πρόσωπα, είπε τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, τους έδωσε ε, μια ε, πλατφόρμα για να μιλήσουν και τους συνάντησε και στη φυλακή. Μετέφερε τα μηνύματά τους στον έξω κόσμο. Ζητώ από εσάς, από εσάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνεχίσετε με αυτή τη δέσμευση και να το κάνετε για όλες σας τις αντιπροσωπείες. Και καμιά αντιπροσωπεία που έχει επαφή με μια κυβέρνηση απολυταρχική που βάζει στη φυλακή τους ακτιβιστές να μην ακούσει τις ξεκάθαρες διεκδικήσεις και απαιτήσει σας να αφαιθούν ελεύθεροι αυτοί οι αντιφρονούντες και να δεσμευτείτε σε επίπεδο κοινοβουλίου με τις εκθέσεις σας ότι θα το πράξετε σε όλη τη διάρκεια. Μάλλον σε όλο το κοινοβούλιο να γίνεται αυτό και όχι μόνο στο πλαίσιο της δικής σας επιτροπής. I can stop here. Μπορώ να σταματήσω εδώ, αλλά πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά, ήδη κάνετε τη διαφορά, αλλά πρέπει από την αρχή με, τη, με τους νέους επιτρόπους να θέσετε το θέμα και να τους στήσετε να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστώ. Τώρα η Κατερίν Ντεντεριάν από την Διεθνή Αμνηστία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω εδώ σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, λόγω της αναθεώρησης του σχεδίου δράσης που, ε, έχει, θα γίνει το επόμενο, διάστημα. Συμμεριζόμαστε και εμείς ε, πολλές από τις ανησυχίες που ακούστηκαν. Για μας η δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να επικεντρώνεται σε αποτελεσματική δράση στη βάση συγκεκριμένων βημάτων τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νέα εργαλεία για την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές καθώς και τα σχέδια δράσης και το στρατηγικό πλαίσιο. Η ύπαρξη αυτών των, των ε, εργαλείων έχει συμβολική σημασία και ε, καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα ε, συστηματικά. Βεβαίως ε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα εργαλεία αυτά με ακόμη πιο φιλόδοξο τρόπο. Σε τρεις τομείς. Πρώτον, εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητα, συνοχή. Μίλησα με συνάδελφο σήμερα το πρωί και είναι ε, εξαιρετικά ενδεικτικό το γεγονός ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο δράσης για το εξωτερικό, ενώ για, το, για ένα εσωτερικό τέτοιο σχέδιο δράσης ακόμη εκρεμεί. Θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν και να διασφαλίσουμε ότι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά τόσο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, θα πρέπει να, γίνει, να γίνουν διπλωματικές ε, κινήσεις. Πολλές φορές υπάρχει σιωπηλή διπλωματία ε, και όχι ε, συγκεκριμένες θέσεις ε, επί, της, επί των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ε, υπάρχει το μέτρο των δημόσιων ανακοινώσεων που πραγματικά έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις όπως αναφέρθηκε. Νομίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να, καταλητικό ρόλο όσον αφορά τη θέση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να γίνουν ορατοί και με αυτό το πνεύμα ε, εκδόθηκε και η δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα για τον Μπουρούντι και τον Κλαβιέρ Γονούμπα. Επίσης, η δημόσια τοποθέτηση θα σημάνει την ε, ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα των ανθρωπίνων διοικηματών, όχι μόνο εδώ σε αυτή την υποεπιτροπή, αλλά και σε περίπτωση, στην περίπτωση συνόδων κορυφής και ε, επισκέψεων υψηλού επίπεδου. Όλα αυτά θα πρέπει να βρεθούν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Τέλος, θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις πραγματικά υλοποιούνται και το επόμενο βήμα, η επόμενη πρόκληση είναι να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, ποια είναι τα συγκριτικά εργαλεία που έχουμε για την ευρωπαϊκή δράση. Για παράδειγμα, ε, συζητήθηκαν ε, στην ΤΡΟΑ πρόσφατα τα, τα εργαλεία, τα benchmarks για αυτόν τον σκοπό. Επίσης, ε, φέτος ε, έγινε και ο διάλογος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικό και υπήρχε και μια τέτοια διάσταση και θα πρέπει να ενισχυθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να ε, καταλήξουμε και σε συγκεκριμένους δείκτες και σε συγκριτικά στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών για το πώς μπορεί να υλοποιηθούν τα σχέδια δράσης και το στρατηγικό πλαίσιο και οι ε, πρωτοβουλίες στα κράτη-μέλη, από τα οποία μπορούν να προκύψουν και βέλτιστες πρακτικές, όπως είδαμε στη Σαουδική ε, Αραβία ή όπως είδαμε σε σχέση με τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων στην Ναμίμπια και στην Ουγκάντα πώς μπορούν αυτά, αυτές οι βελτιές πρακτικές να εφαρμοστούν και σε άλλες περιπτώσεις και για να κλείσω πώς μπορούμε να απαντήσουμε στην πράξη σε αυτό το ζήτημα όσον αφορά την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια σε ολόκληρο τον κόσμο φέτος έχουμε μπροστά μας την 30η ε, επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των ε, βασανιστήριων. Είναι μια ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση και ρόλο και να τοποθετηθεί κατά των βασανιστήριων. Για παράδειγμα, μπορούμε να ε, επικεντρωθούμε στην παρακολούθηση των βασανιστήριων σε τρίτες χώρες και να τις δημοσιεύσουμε ώστε να μπορέσουν και οι εμπλεκόμενοι φορείς να ανταλλάξουν απόψεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι κάνουν σχετικά με την κακομεταχείριση και, τον, ε, και τα βασανιστήρια. Θα μπορούσε να είναι και ένα μόνιμο στοιχείο αυτό στον ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες. Έτσι θα μπορούσαν τα βασανιστήρια να γίνουν ένα ε, ζήτημα που θα περιβάλλεται από πολιτική ευαισθησία. Μιλάμε και για τις εξαφανείς ανθρώπων. Αυτό το κάνουμε, ε, αλλά δεν μιλάμε ποτέ για τα βασανιστήρια. Επίσης, για την συνοχή μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής δράσης, όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επικυρώσουν την OPCAT όπως ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζητά αυτό από τρίτες χώρες. Επίσης τα κράτη-μέλη μπορούν να ε, τιμήσουν αυτήν την ε, επέτειο των 30 ε, ετών εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές για την ε, υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να βασιστεί στις δικές του, στα δικά του ψηφίσματα τις περσινής χρονιές προκειμένου να πιέσει για ακόμη μεγαλύτερη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση φέτο. Κάποιε ιδέε είναι αυτέ για το πώ μπορούν οι στόχοι, οι δεσμεύσει να ε, υλοποιηθούν. Και βεβαίω θα παρακολουθήσουμε από κοντά και την ε, συζήτηση που θα γίνει στο το επόμενο διάστημα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ε, ευχαριστούμε και τους τέσσερις, η ε, έχει λάβει μια, ε, μεγάλη, έναν μεγάλο κατάλογο ε, με ιδέες από το δίκτυό σας, τον οποίο βεβαίως θα λάβουμε υπόψη. Όπως είπα, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Παντζέρη, που είναι ο εισηγητής της ετήσιας έκθεσης και στη συνέχεια στα μέλη. Πείτε μου σας παρακαλώ αν θέλετε να λάβετε το λόγο και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Σέρι από την EAS και αν έχουμε χρόνο τότε θα δώσω το λόγο ξανά στους ομιλητές ή για, το, για τοποθετήσεις ή για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. Σας ευχαριστώ. Θα πρέπει καταρχήν να πω πως ευχαριστώ όλους ε, για τη συμβολή σας. Δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω ωστόσο ότι τους επόμενους μήνες θα χρειαστεί να κάνουμε πολύ πολύ σοβαρή και εις βάθος ε, δουλειά. Έχουμε μπροστά μας ε, πολύ σοβαρό έργο. Και δεν ξέρω αν θα είμαστε σε θέση να, δώσουμε, να κάνουμε μάλλον μία νέα αρχή, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Εγώ πιστεύω και συμφωνώ με τα λόγια της κυρίας Σαλ ότι δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να θεωρούνται, δηλαδή θα εργαστώ σε τέσσερις άξονες βασικά. Καταρχήν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα κάθε δράση ε, στην οποία προφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ενισχύουν και ενισχύονται βέβαια και τα δικά σας λόγια ότι είμαι υπέρ του να είναι ένα οριζόντιο θέμα, να διέπει δηλαδή και όλα τα άλλα. Και ωστόσο θα πρέπει να έχουμε και τον απαραίτητο ρεαλισμό και να πούμε ότι δεν θα είναι απλό αυτό γιατί υπάρχουν χώρες αλλά και άτομα που πιστεύουν πως τα δικαιώματα είναι κάτι είναι, κοστίζουν και ότι δεν χρειάζονται και σε τίποτα. Και το βλέπουμε με διάφορες εκφράσεις. Σήμερα το πρωί, α πούμε, συζητήσαμε για ένα σημαντικό θέμα, δηλαδή τα δικαιώματα των εργαζομένων στον κόσμο. Ε, για να δώσουμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα. Δεν θα είναι απλό λοιπόν, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε, να το προσπαθήσουμε. Εγώ πιστεύω και θα το γράψουμε αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε κοινή δουλειά με όλε τι επιτροπέ ε, του Κοινοβουλίου τοποθετώντας στο επίκεντρο τρία-τέσσερα θέματα που θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων. Γιατί θεωρώ πως είναι βασικό αίτιο για την έλλειψη δικαιωμάτων. Το άλλο θέμα είναι αυτό που τελευταία αναφέρθηκε, δηλαδή καταπολέμηση των βασανιστήριων και των κακής μεταχείρισης. Σκέφτομαι επίσης το θέμα ότι βρισκόμαστε στην ε, κυοφορία της ε, Διατλαντικής Εμπορικής Συμφωνίας. από το θέμα του να είναι τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κομμάτι αναπόσπαστο των εμπορικών συμφωνιών στις οποίες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες εκτός Ένωσης και τέλος το θέμα της στήριξης στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού. Θα πρέπει πολύ να σκεφτούμε για τις διάφορες, ε, τα διάφορα αυτά θέματα και πρέπει να μας απασχολήσουν διότι μεταξύ άλλων ίσως πρέπει να ερμηνεύσουμε τις πολιτικές που ασκούνται, για παράδειγμα, την αρχή της, του More for More, που δεν ξέρω τι αποτελέσματα είχε στις διάφορες χώρες. Πρώτο πεδίο λοιπόν. Δεύτερο πεδίο είναι αυτό των μεμονωμένων χωρών, των, της παρέμβασης αναχώρα. Όπως γνωρίζετε κάλλιστα, χρησιμοποιούμε ψηφίσματα και τα κατεπήγοντα θέματα, αλλά εδώ πιστεύω θα πρέπει να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που είναι η κατάσταση πρόοδου των μεμονωμένων θεμάτων, διότι στην πράξη λίγα γνωρίζουμε. Ε, το έχουμε κάνει. Ε, αλλά πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε κάτι πετύχει ή όχι, γιατί εφόσον δεν είχαμε αποτελέσματα θα πρέπει να επανέλθουμε. Ε, αν τα έχουμε πετύχει είναι ένα σημαντικό στοιχείο καλής πρακτικής που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για άλλες υποθέσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ορατή και διαφανής η διαδικασία για τις διάφορες ε, πολιτικές. Θα ήταν ίσως σκόπιμο, αλλά είναι και αυτό δύσκολο να έχουμε περισσότερη ευελιξία από πλευρά του Κοινοβουλίου για τα μεμονωμένα προβλήματα. Από τη συζήτηση που μόλις κάναμε για τον Μπαχρέιν, ε, θα έλεγα ότι δεν θα ήταν δύσκολο να πάρει κανείς μια άμεση θέση Άμεσα τώρα να πούμε ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δημοκρατικές τις εκλογές εφόσον όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν στη φυλακή. Ε, αυτό μπορούμε κάλλιστα να το κάνουμε χωρίς να περιμένουμε να μας δώσει το OK, το επίσημο, να μας το δώσουν όλες, όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Τέλος, στα δυο άλλο πλαίσια, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν προθεσμίες σε στρατηγικό επίπεδο γιατί εκπνέει το 2000, εκπνέουν κάποια πράγματα το 2014 και είναι σημαντικό να συμβάλλουμε στον ορισμό του στρατηγικού ε, πλάνου για το 2015. Αυτό σημαίνει στην ουσία για μένα να απαιτήσουμε πέρα από το Κοινοβούλιο τις διάφορες ΜΚΟ ε, και τους διάφορους οργανισμούς να, αποτελέσουν, να, να, συμμετέχουν στον ορισμό αυτού του στρατηγικού σχεδίου και επίσης να πω πως θεωρώ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική μάλιστα, τη δουλειά που έχει κάνει η ειδική εκπρόσωπο, ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σταύρος Λαμπρινίδης, που κατά τη γνώμη μου όχι μόνο θα πρέπει να στηριχθεί, αλλά και να ενισχυθεί η δουλειά του, ακριβώ γιατί πρέπει να παρεμβαίνει σε μεμονωμένε χώρε. Τέλο, τέταρτο πεδίο είναι η εξωτερική πολιτική. Ήδη είχα την ευκαιρία για ανεπίσημη συνομιλία με την μελλοντική, είπατε, εκπρόσωπη, εκπρόσωπο που θα ε, εγκριθεί μάλλον μέσα στις επόμενες εβδομάδες με τη Φεντερίκα Μογκερίνη. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να συνοδεύει τη δράση τόσο τη εξωτερική μα πολιτική γενικότερα όσο και τη άλλη πτυχή τη εξωτερική πολιτική που είναι η πολιτική γυρνίασης και είναι και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο. Και αυτό είχα την ευκαιρία να το συζητήσω με την υποψήφια είπα εκπρόσωπο και τον Επίτροπο Άρμστερ για την ε, ε, πολιτική γειτονίας. Τέλος να κλείσω και Στη διάρκεια λοιπόν ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης θα έχουμε μια συζήτηση και επαφή με όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις ενώσεις τους. Ε, ε, αυτά έχω να πω για σήμερα ως πρώτο, στοιχεία για την ετήσια έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Παντζέρη. Κυρία Βερζιά, ευχαριστώ. Γρήγορα, γρήγορα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω όλες φιλικό το πάνελ. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό αυτά το οποία αναφέρετε. Είχα την ευκαιρία να το πω σε κάθε μία από εσάς ή οργανώσεις σας τουλάχιστον και παραμένω πιστή στα λόγια μου. Αλλά δεν έχω ικανοποιηθεί επαρκώς. Ίσως γιατί σας πιέζει ο χρόνος και έπρεπε να μείνετε έτσι σε κάποιες γενικότητες ίσως, αλλά νομίζω ότι θα χρειαζόταν να μας δώσετε παραδείγματα, ιδίως σε σχέση με την έκθεση της Κομισιόν, για κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν, γιατί νομίζω ότι όταν ε, αναφέρουμε παραδείγματα για κάποιες ε, θεματικές, ε, είμαστε πιο ισχυροί. Αλλιώς, αν παραμείνουμε γενικοί, δεν δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος Παντσέρη. Πιστεύω ότι επανακαθορισμός στρατηγικού πλαισίου είναι σημαντικό θέμα και ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε και με τέτοιες συναντήσεις, κάποια σημεία στήριξης. Δεν ξέρω τώρα σε ποια συνάντηση, πάντως κάπου είχε γίνει λόγος ε, για την ανάγκη, πώς να το πω τώρα, το στρατηγικό πλαίσιο να είναι διαφορετικό αναχώρα Και οι μη κοινωνικέ οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν γιατί γνωρίζουν την κατάσταση. Είναι ένα σημείο λοιπόν επαφής εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τα κατεπήγοντα κυρίως και νομίζω ότι μπορούμε από κοινού να επεξεργαστούμε αυτά τα θέματα που είναι σημαντικά κατ' εμέ. Έχουμε πολύ καλή δουλειά να κάνουμε. Είναι καλό εργαλείο το στρατηγικό πλαίσιο 2012, αλλά πρέπει να εργαστούμε τώρα και έχετε κι εσείς την πρόθεση από ό,τι φαίνεται να το κάνετε για το μέλλον. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Αν όχι, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις και σχόλια. Για την κυρία Χάλ, που είπε ότι είναι καλό να έχουμε τακτικές ανταλλαγές ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πράγματι το κάναμε αυτό κατά το παρελθόν, φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ήταν όμως έτος εκλογών το 2014, οπότε το 2015 φαντάζομαι θα συνεχίσουμε την πρακτική αυτή. Δεν θέλω να ε, συζητήσω πάνω σε όλες τις ε, συστάσεις που έγιναν. Για την κυρία Ντουσεπούλκρε, για την ποιότητα των μελετών αντικτύπου. Μας απασχολεί και εμάς αυτό το θέμα και μόλις σήμερα το πρωί είχαμε μια ακρόαση και ασχοληθήκαμε ακριβώ με αυτό. Την κακή αξιολόγηση της κατάστασης στη Βιρμανία. Νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα θα είναι στις εργασίες μας και αυτό ένα θέμα και το ότι πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και των ειρηνικών ακτιβιστών. Ε, μας κάνατε μια έντονη έκκληση. Θα το κάνουμε, αλλά ξέρετε αυτό είναι μια συνεχιζόμενη δουλειά. Αναφερθήκατε στην κυρία Γιούνος από το Αζερμπαϊτζάν και στον κύριο Πιέρ, τώρα το όνομά του, το επιθετό από τον Μπουρούντι δεν το θυμάμαι να το πω, αλλά εγκρίναμε για αυτού τους δύο που αναφέρατε ψηφίσματα στο Κοινοβούλιο. Να κάνω και ένα ερώτημα προς όλες σας ίσως. Ξεκινάμε από την αρχή, έχουμε μια νέα νομοθετική εξουσία, έχουμε νέους ε, συναντέλφους, πολλούς στον αριθμό και αν δείτε τα πολιτικά προγράμματα ε, πολλών κομμάτων, ε, πολλών συναδέλφων, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες πολιτικές. Κάποιοι, παραδείγματο χάρη, είναι υπέρ της θανατικής ποινής ε, ή για εισαγωγή της θανατικής ποινής. Ε, κάποια γαλλικά κόμματα, ιδίως το εθνικό μέτωπο, το Front National, αυτό το περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του, το εκλογικό. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό και εσείς από την πλευρά των ανθρωπίνων κοιμάτων να παρακολουθείτε λίγο και το τι λένε τα κόμματα στα προγράμματά τους. Επίσης θα ήθελα γιατί το είπε και ο κ. Παντσέρη. Έχουμε τις ακροάσει ε, των επιτρόπων. Έχουμε τον κύριο Χάν στην ΑΦΕΤ και με την κυρία Μογκερίνη. Και έχω ένα ερώτημα που δεν ξέρω τι απάντηση μπορεί να έχει. Αυτή η νέα δομή που συγκροτεί ο Γιούνκερ. Πώς έχει αυτή η δομή, θα ωφελήσει με αυτή την εγκάρσια προοπτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή θα περιπλέξει την κατάσταση. Αν μπορείτε να απαντήσετε. Γιατί με απασχολεί και εμένα αυτό το ερώτημα. Να ακούσουμε τώρα τον κύριο Σέρι από την ΙΕΔ, την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ευχαριστώ. Κάποιε παρατηρήσεις για όσα ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα, σε προσωπική βάση επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω Νομίζω ότι γνωρίζω όλους ε, τους συμμετέχοντες του πάνελ γιατί έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ε, στο παρελθόν. Ένα χρόνο δουλεύω εγώ και ήδη είχα πολλές φορές την ευκαιρία να ε, συζητήσουμε με το δίκτυο και με την κοινωνία των πολιτών. Είναι τμήμα της δουλειάς μας λοιπόν. Είναι, ε, προσπαθούμε βεβαίως να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας αλλά και να συλλέξουμε όσο περισσότερα στοιχεία ακριβώς για να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις και την κριτική που έρχεται από την κοινωνία των πολιτών. Πολύ θετικό λοιπόν αυτό. Τώρα, για τα ζητήματα που τέθηκαν, για πρώτη φορά ήταν συστάσεις προς το Κοινοβούλιο, ε, ε, αλλά υπάρχουν συστάσεις βεβαίως και για τη δική μας δράση, για τα σχέδια δράσης, κάποιες αδυναμίες που αναφέρθηκαν και που τονίστηκαν σε κάποια ζητήματα συμφωνούμε απολύτως. Πρώτα και κύρια στο γεγονός ότι συμμεριζόμαστε και εμείς την άποψη ότι το στρατηγικό πλάσιο και το σχέδιο δράσης ήταν τουλάχιστον μια επιτυχημένη προσπάθεια, μια κοινή προσπάθεια για να δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα στο ζήτημα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια προσπάθεια για να ε, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Κάποιες φορές ήμασταν επιτυχημένοι, κάποιες φορές όχι και τόσο, αλλά πάντως ε, σε κάθε περίπτωση κάναμε προσπάθειες και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να κάνουμε και βεβαίως επεξεργαζόμαστε και ένα νέο σχέδιο δράσης. Ε, μπορώ να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Επίσης, σημείωσα ε, πολλά ζητήματα που τέθηκαν και στα οποία νομίζω ότι συμφωνούμε τέθηκε το ζήτημα των, ε, της εκτίμησης ε, κινδύνου, ε, της συνοχής των πολιτικών μας. Όλα αυτά βεβαίως είναι ζητήματα που χρειάζεται να κάνουμε ακόμη περισσότερα σε πολλές περιπτώσεις και βεβαίως και στο μέλλον και βεβαίως θα ε, κατανείμουμε και πολλούς πόρους και θα κάνουμε πολλές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει και το ζήτημα της συνοχής της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης. Είναι μια συζήτηση που σίγουρα θα πρέπει να γίνει ε, και στο μέλλον θα γίνουν προσπάθειες και προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα ότι έχουμε αποτύχει στο να απελευθερώσουμε ανθρώπους. Βεβαίως μπορούμε να βελτιώσουμε τις δράσεις μας να εντοπίσουμε και κάποιες αδυναμίες, αλλά συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι πρόκειται για μια ε, εργασία που βρίσκεται σε εξήλυξη. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναλάβει πάρα πολλές δραστηριότητες και εμείς σε καθημερινή βάση συνεργαζόμαστε με αντιπροσωπείες που εργάζονται ακριβώς για αυτόν τον σκοπό, για να απελευθερώσουν κόσμο, πολλές φορές ε, ίσως ε, δεν είμαστε ορατοί, κάποιες φορές ίσως δεν πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα ορατοί, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδεχομένως πράγματι να μην έχουμε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι μας, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ιστορίες επιτυχίας που πολλές φορές μπορεί να μην έχουν γίνει δημόσιες. Για παράδειγμα στην περίπτωση του, Μπαχρο... του Μπαχρέιν, που ο συνάδελφός μου ε, με διαβεβαιώνει ε, ότι έχετε κάνει κι εσείς πολλά ψηφίσματα, πολλές ε, ανακοινώσεις. Είναι πάλι ένα ζήτημα ερμηνείας, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε άδικοι λέγοντας ότι έχουμε αποτύχει σε όλα αυτά. Τώρα για το ζήτημα των ακτιβιστών, ε, αυτά για, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το άλλο ζήτημα που ήθελα να αναφέρω, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, γιατί στην τελευταία συνεδρίαση της υποτροπής Ντρουά είχε συζητηθεί με τον Σίλβιο Κολζάτο, με τον Διευθυντή, το μέλλον του σχεδίου δράσης. Μπορώ να σας πω πάντως ότι, και να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή ε, εργαζόμαστε πάνω σε μια αξιολόγηση της δράσης μας που θα είναι η βάση ε, επί της οποίας θα χαράξουμε το νέο σχέδιο δράσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συζήτηση με την Κομισιόν, με τους συναδέλφους από την Κομισιόν και θα γίνει και συζήτηση επ' αυτού στις αρχές Οκτωβρίου και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε και βεβαίως με τα χαράς θα ε, κάνουμε και συναντήσεις με το δίκτυο και με την κοινωνία των πολιτών τον Οκτώβριο, αν και εσείς συμφωνείτε. Ίσως να χρειάζεται να επαναλάβω ότι είμαστε ε, απολύτως ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση με το Κοινοβούλιο στο μέλλον. Το Κοινοβούλιο είναι ο βασικός μας εταίρος όσον αφορά την ε, ε, κατάρτιση αυτού του νέου σχεδίου δράσης και κύριε Παντσέρη άκουσα και την, ε, τις δικές σας απόψεις, την, ε, τον τρόπο με τον οποίο περιγράψατε δική σας έκθεση. Με τα χαράς βεβαίως θα ε, συνεργαστούμε και μαζί σας αν και εσείς συμφωνείτε και αν χρειάζεστε βεβαίως οποιαδήποτε από την πλευρά μας υποστήριξη στις δικές σας εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε έχουμε μείνει, ναι, έχει μείνει λίγος χρόνος να ξεκινήσω τώρα ανάποδα και να αν μπορούσα να σας ζητήσω να απαντήσετε για τις συστάσεις. Ξεκινάω με την κυρία Τεντέριαν. Ήταν πολλά τα σχόλια, δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε όλα. Ευχαριστώ πάντως για το σχόλιο της κυρίας Βερζά για το ότι χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Ένα στοιχείο, μια περίπτωση είναι η περίπτωση του κύριου Κλαβιέ Εκεί πράγματι υπήρχαν Υπήρχαν δηλώσεις επιτόπου για, τον, ε, για το συγκεκριμένο άνθρωπο και βοήθησε πολύ. Δυστυχώς όμως αυτά τα, τα ψηφίσματα δεν αναφέρονταν ποτέ σε εκείνον ως ε, υπερασπιστή των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης δεν, αναφέρ, δεν ανέφεραν τις διεθνείς ε, δεσμεύσεις του Μπαχρέιν, δεν ανέφεραν τις ε, υποχρεώσεις. Χρειάζεται να κάνουμε πολλή δουλειά βεβαίως. Κατανοώ ότι ε, θα πρέπει να γίνει δουλειά και επιτόπου και βεβαίως χαιρετίζουμε το ψήφισμα του, ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Τη χαιρέτησε βεβαίως και η κοινωνία των πολιτών στο Μπαχρέιν. Οπότε σας ευχαριστούμε βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος εντός των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την απελευθέρωσή του. Το δεύτερο σχόλιο. Ευχαριστώ για το σχόλιο βεβαίως για το σχέδιο δράσης και για τα συγκριτικά στοιχεία της, πρακ... της Στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ντρουά αναφέρθηκε ότι το 2013 υπήρξαν 96 ε, δηλώσεις στις Βρυξέλλες και 36 δηλώσεις σε τοπικό επίπεδο όπου αναφέρονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ο λόγος για τον οποίο ζητούμε αυτήν την σαφήνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι κατά πόσο ήταν σαφές τελικά το μήνυμα αυτών των ανακοινώσεων και ποιο ήταν και το αποτέλεσμα αυτών των ε, ανακοινώσεων. Ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό για το μέλλον να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Λότε Λάιχτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε να ξέρετε για την κατάσταση σε μια χώρα, τι είδους κυβέρνηση έχει, πώς ε, μεταχειρίζεται το λαό της. Μην βλέπετε, μάλλον κοιτάξτε πρώτα απ' όλα στις φυλακές και αν εκεί υπάρχουν ειρηνικοί ακτιβιστές κάτι πολύ λάθος υπάρχει σε αυτή τη χώρα και από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε και αυτό πρέπει να είναι κομμάτι του διαλόγου που έχετε με την οποιαδήποτε τέτοια χώρα και πρέπει να είναι και δική σας φιλοδοξία για να αλλάξει η κατάσταση και να επηρεάσετε το πώς μεταχειρίζεται το λαό της. Πρέπει να βγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη φυλακή, αυτοί οι οποίοι θέλουν ειρηνικά να διαδηλώσουν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Η αλλαγή πάντοτε έρχεται εκ των ένδων. Δεν έρχεται από εσά, εσείς μπορείτε να βοηθήσετε και σίγουρα να τονίζετε αρχές βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Όμως, οι άνθρωποι είναι αυτοί που επηρεάζουν τις αλλαγές και όταν είναι στη φυλακή σταματάει η ειρηνική αλλαγή. Άρα, η φιλοδοξία σας και προτεραιότητά σας πρέπει να είναι προσπίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα κάνετε τη διαφορά να πετύχετε. Άρα θα πρέπει να βάλουμε πιο ψηλά τον πύχη της φιλοδοξίας για να βγουν πιο πολλοί άνθρωποι από τη φυλακή. Δεν μπορώ να φανταστώ μια πιο καλή κληρονομιά ε, για τη νέα υπάτη εκπρόσωπη και για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες να πετύχετε να είναι έξω από τις φυλακές οι ειρηνικοί διαδηλωτές, ακτιβιστές υπέρ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα κληροδότημα τεράστιο. Και ακούσαμε και για τον Μπαχρέιν. Έχουμε το... βασικό ε, παράδειγμα ε, με τον Αμπτούλ Χαντί Αλκαβάγουα που είναι στη φυλακή και είναι και αυτός ένας ε, πολίτης που δεν μπορεί να να βγει από τη φυλακή χωρί τη δική σας βοήθεια. Άμα δεν βάλετε όλο σα το βάρος αυτή την προσπάθεια, πώς θα πείσετε ότι έχετε πραγματική ε, βούληση να βοηθήσετε τους παράγοντες ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σας ζητούμε λοιπόν να δώσετε, να έχετε ένα θεματολόγιο για, την, για το δικαίωμα των ανθρώπων να ασκούν τα δικαιώματά τους. Σε ό,τι αφορά το στρατηγικό πλαίσιο, Δεν νομίζω ότι αξίζει να δαπανιστεί πολλή χρόνο για την εκπόνηση ενό νέου στρατηγικού πλαίσιο. Θέλουμε να δούμε τη νέα εποχή εφαρμογή αυτού του στρατηγικού πλαίσιου. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο. Είναι μια δέσμευση που προήλθε από το ότι ΜΚΟ, ευρωπαϊκοί θεσμοί, ε, κράτη-μέλη συνεργάστηκαν μεταξύ τους και είναι σημαντικό όλοι να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Εμείς ε, αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τον πολύ σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου και πριν και τώρα και σας παρακαλούμε να κάνετε ακόμη περισσότερα. Σε ό,τι αφορά τις ε, στρατηγικές αναχώρα, έχει ζητηθεί πολλάκις να μην είναι μυστικά αυτά τα έγγραφα και αυτές οι εκκλήσεις προέρχονται και από τα κράτη-μέλη. Άρα πρέπει να ασκηθεί πίεση από το Κοινοβούλιο ώστε τουλάχιστον οι βασικές ανησυχίες και μελήματα να κοινοποιηθούν, να δημοσιοποιηθούν, ώστε να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε την αξιολόγηση που θέλουμε να γίνει. Μέρος του προβλήματος είναι ότι όσοι συνεισφέρουμε σε αυτές τις στρατηγικές των χωρών, μένουμε στο σκοτάδι. Και μόνο άμα διαρρεύσουν τα έγγραφα βλέπουμε αν οι συστάσεις μας έχουν συμπεριληφθεί ή όχι και αν Γίνεται λόγος για αυτές στις συναντήσεις των, υπαλλή, των ε, αξιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εκπροσώπους τρίτων χωρών. Κάτι που λείπει είναι η φιλοδοξία τελικά. Να βγουν από τη φυλακή οι ακτιβιστέ, οι υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις στρατηγικέ των χωρών αυτή πρέπει να είναι μια προτεραιότητα σημαντική με μια τρίτη χώρα που έχει τέτοιους ανθρώπου στι φυλακέ τη. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα η Γκέλ Ντουσεπούλκρα. Ευχαριστώ. Σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, θα ήθελα να σας δώσω τρεις προθεσμίες. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία αναθεώρησης των κατευθυντήρων γραμμών για τις μελέτες ε, επιπτώσεων και ανησυχούμε για το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά η κατευθυντήρια γραμμή που εκδόθηκε από την Κομισιόν το 2011 για το πώς αντιμετωπίζουν, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις διαβουλεύσεις λοιπόν δεν υπάρχει καμία αναφορά όσον αφορά ε, τα βήματα που θα γίνουν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, η δεύτερη προθεσμία, η DigiTrade, βρίσκεται επίσης στη διαδικασία αναθεώρησης της ε, δικής της ε, ε, στρατηγικής. Η τρίτη κατευθυντήρια γραμμή, για παράδειγμα, αφορά την σύναψη συμβάσεων εμπορικού χαρακτήρα ή για, συμβάσεων επενδύσεων. Έχουμε για παράδειγμα το, την περίπτωση του Βιετνάμ που έχει σχεδόν κλείσει και ε, ενημερώσαμε τον συνήγορο του ε, πολίτη ότι δεν υπάρχει μελέτη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επειδή λοιπόν το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει αυτές τις μελέτες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ, ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει και το ζήτημα αυτό. Αυτά όσον αφορά τη μελέτη ε, επιπτώσεων. Τώρα, για συγκεκριμένα παραδείγματα που ζητήθηκαν. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει και πιέζει τις χώρες να ε, επικυρώσουν ε, την σύμβαση της Ρώμης. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία γιατί ακούσαμε στους, διαβάσαμε στον ε, ε τύπο ορισμένες ε, ανακοινώσεις. Τώρα για τη στρατηγική πρέπει να σας πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα συγκλίνουν ώστε να υποστηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, στη Βυρμανία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επικυρώνει συμφωνίες με το εμπορικό επιμελητήριο, αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στη συμφωνία αυτή. Οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αναφορά στις κατευθύνες γραμμές του ΟΗΕ. Θεωρούμε επίσης ότι το γεγονός ότι η νέα ύπατη εκπρόσωπος θα ε, επισκέπτεται και θα συνεργάζεται ε, συχνά με διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα βοηθήσει τόσο στο συντονισμό όσο και στη συνοχή των πολιτικών. Συμφωνήσαμε επίσης για τις νέες αρμοδιότητες που μπορεί να αναλάβει ο κύριος Τίμερμανς. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπιστούν τα βασικά προβλήματα. Για παράδειγμα, πιστεύω... Ε, συγγνώμη, ε, ε, ένα τελευταίο πράγμα. Πρέπει να γίνει να σιγουρευτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα γίνει σεβαστή σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ε, αν έχετε και άλλες συστάσεις θα χαρούμε πολύ να μας τις στείλετε και γραπτός. Και τέλος για Χάιντ pick Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι πιο ωραία όταν είναι καταγεγραμμένα. Πολλά από όλα αυτά που λέει και γράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνονται πολύ θετικά, όμως θα πρέπει να γίνουν και εκκλήσεις για εφαρμογή. Ε, κύριος ε, Τίμερμανς έχει θα, πρέπει ναι, να ε, ασχοληθεί με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυρία Μογκερίνη, με πάρα πολλά θέματα. Θα θέλαμε και το εμπόριο σίγουρα να περιλαμβάνεται εκεί και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά πράξη, γι' αυτά προσβλέπουμε στο Κοινοβούλιο. Γιατί άλλο είναι τα όσα γράφονται και άλλο είναι τι γίνεται στην πράξη. Προσβλέπουμε λοιπόν σε στενή συνεργασία μαζί σας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα τεθούν και όλα σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ και εμείς σας ευχαριστούμε και τώρα έχω ένα αίτημα από τον κύριο Φέρη για ένα λεπτό. Ναι, πολύ σύντομα να δώσω μια τεχνοκριτικού τύπου λεπτομέρεια. Έχουμε διάφορα έγγραφα, ένα στρατηγικό πλαίσιο και έχουμε και το πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει καμιά διάθεση να αλλάξει το στρατηγικό πλαίσιο το ίδιο. Είναι ένα γενικό πλαίσιο αυτό, είναι πολύ καλό, αλλά αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για την ανανέωση, μάλλον αξιολόγηση και ανανέωση του προγράμματος δράσης, που είναι πιο συγκεκριμένο, πιο πρακτικό έγγραφο γιατί εστιάζει την προσοχή σε συγκεκριμένε δράσεις. Κάποια πράγματα έχουν ήδη γίνει, κάποια θα πρέπει να ανανεωθούν κτλ. Αυτά για να σας διευκρινίσω, να είμαστε πιο ακριβεί. Αλλά βέβαια το πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε είναι ότι η δουλειά που έχουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει τελικά να εγκριθεί και από την νέα ύπατη εκπρόσωπο. Ό,τι και αν λέμε εμεί εδώ, ναι, είναι η καθημερινή μα δουλειά, σε αυτά στοχεύουμε, αλλά βέβαια θα πρέπει η τελική απόφαση να ληφθεί από την κυρία Μογκερίνη. Και να ευχαριστήσω και πάλι όλες τις ομελέτριες που ήταν σήμερα εδώ και θα είστε μαζί μας και τα επόμενα πέντε χρόνια. Και τώρα παρακαλώ τους υπηρογνώμονες στο επόμενο πάνελ να έρθουν. Ανταλλαγή απόψεων για τα βασανιστήρια και τη θανατική ποινή. Um, actually, we start this exchange um, with a message from. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ανταλλαγή με ένα μήνυμα του Φεντερίκο Μέγερ. Τεχνικά μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά σας, οι διερμηνείς δεν θα το μεταφράσουν.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 Ευχαριστώ εγώ, κύριε Φεντερίκο Μάγιορ. Ο συνικός Διευθυντής της UNESCO με πολύ ε, ε, ολιστική προσέγγιση για τον πολιτισμό και την ειρήνη, είναι τώρα πρόεδρο τη Διεθνούς Επιτροπή κατά τη Θανατική ποινή Και έχουμε συστάσεις από τον ίδιο οργανισμό, τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Σούντα Βίβο Καβαλιέρ. Ο Φεντερίκο Μέιερ ήταν στις Βρυξέλλες πέρυσι που έκανε μια πολύ έντονη έκκληση να συνεχίσουμε στην Ένωση και στο Κοινοβούλιο να εστιάζουμε στην κατάργηση της θανατικής ποινή. Στα διεθνή φόρα βεβαίως βλέπετε ότι είναι απόλυτα απαραίτητο να πιέζουμε διαρκώς για να προωθούμε αυτό το θέμα. Πριν να δώσω το λόγο στους συμπειρογνώμονες θα ήθελα να διαβάσω τα όσα προετοιμάστηκαν από την γραμματεία μας για να μας θυμίσουν ότι βέβαια συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που, είναι, που, έχουν ε, καταδικαστεί στη θανατική ποινή για να δούμε αν υπάρχει κάποια τάση. Το 2013 ο αριθμός των εκτελέσεων αυξήθηκε κατά 50% σχεδόν σε σχέση με το 2012. Ακόμα και αν δεν μετρήσουμε την Κίνα, γιατί δεν έχουμε από εκεί επίσημα στοιχεία, γιατί είναι κρατικό μυστικό, ε, χωρίς την Κίνα 778 άνθρωποι εκτελέστηκαν στον κόσμο. 80% σε τρεις χώρες μόνο. Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σαφώς μειονέκτημα λοιπόν όταν ε, συγκρίνουμε αυτά τα νούμερα αλλά μπορούμε να δούμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου που έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής. Και στις 10 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, και φέτος είναι η 12η Διεθνής ημέρα κατά της θανατικής ποινής, πιστεύω πως αυτή τη φορά εστιάζεται περισσότερο στους ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί και που αντιμετωπίζουν την θανατική ποινή που ψυχικά είναι άρρωστοι. Έχουμε καλέσει τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Επιτροπής κατά της, ε, την Γενική Γραμματέα, την κυρία Καβαλιέ, τον κύριο Ντέιβιτ Nichols από την Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας και νομίζω πως θα μας ενημερώσετε για τη θανατική ποινή, αλλά και για τον κανονισμό περί εργα... εργαλείων βασανιστήριων του ΟΗΕ γιατί, όπως ακούσαμε στην προηγούμενο μας θέμα, προετοιμάζεται ένας νέος κανονισμός. Νομίζω πως εδώ ε, συνεχίζουμε τον αγώνα. Ε, δεν έχουμε ε, ακόμα αποφασίσει ποια επιτροπή θα ασχολείται με το θέμα και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να προετοιμάσουμε το περιεχόμενο μιας γνωμοδότησης. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακόμα ποια επιτροπή θα την κάνει και η κυρία Φώ που είναι σήμερα από το πρωί εδώ από την ε, μη κυβερνητική Rebrief, που είναι στρατηγική ε, διευθύντρια της ομάδας για την θανατική ποινή και είναι υπεύθυνη για την εκστρατεία στα, ε, για stop στο πρόγραμμα θανατηφόρων ενέσεων είναι μικρή αυτή η ΜΚΙΟ σε σχέση με άλλες τεράστιες ε, ε, οργανώσεις, αλλά έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στις διεθνείς συνεργασίες όσον αφορά την πώληση, την εξαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση. Για παράδειγμα, στη χώρα μου, τη Γερμανία, νομίζω εσείς και μερικοί ακόμα μαζί βοηθήσατε έτσι ώστε για το Φραζένιος Κέρ ε, να σταματήσει να ε, κάνει αυτή τη ε, διαδικασία και, το ίδιο δεν βοηθήσατε για να σταματήσει, να καταργηθεί μάλλον η θανατική ποινή σε όλες τις πολιτείες της, των ΙΠΑ. Σε κυρία Σούντα Καβαλιέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε για να παραστούμε εδώ στην Συνέδριση που Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Συνεχίζοντας στο πνεύμα της ομιλίας του Προέδρου μας, του κύριου Μαγιόρ, πιστεύω και εγώ ότι οι βουλευτές είναι εξαιρετικά σημαντικοί στον αγώνα κατά της ε, θανατικής ποινής. Μια ε, ε, μεγαλύτερη δραστηριοποίηση θα μπορούσε να, να ε, ασκήσει πιέσεις για την κατάργηση ε, της θανατικής ποινής. Ε, πέρσι έγινε και μια αντίστοιχη ε, εκδήλωση, μια συνάντηση με ε, βουλευτές από 11 χώρες για να συζητηθεί η, καταδίκη, κατάργηση της θατικής ποινής ε, από την Αυστραλία, το, την Ιαπωνία, τον Μπαχρέιν, την Ορδανία, το Πακιστάν, το Σουρινάμ, το Περού και την ε, Ζάμπια. Το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών μεταξύ των ε, βουλευτών, βουλευτής από το Σουρινάμ δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει δράση για την κατάργηση της θανατικής ποινής και ως συνέχεια αυτής της συζήτησης ε, διοργανώθηκε μία αποστολή του ICDP στο Σουρινάμ και μία από, ένα από τα μέλη, η κυρία Ντρέισφος, που ήταν ε, βουλευτής και ε, μέλος αυτής της αποστολής, έδωσε την ε, βοήθειά της ε, σε άλλους βουλευτές στο Σουρινάμ. Στο τέλος αυτής της αποστολής δηλώθηκε στους τύπες, στον τύπο ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Σουρινάμ θα αναλάβει ε, δράση προς την κατάργηση της θανατικής ποινής. Αυτή τη στιγμή γίνεται αναθεώρηση του ποινικού κώδικα και δεν γίνεται καμία αναφορά στην θανατική ποινή. Επίσης ε, διοργανώνονται σεμινάρια την, ε, τον επόμενο χρόνο στο Σουρινάμ προκειμένου να επικυρωθεί το ε, δεύτερο πρωτόκολλο. Και υπάρχει και υπεύθυνο για αυτήν την προσπάθεια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό, διότι σήμερα, ε, φέτος, ε, συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υιοθέτηση του πρωτοκόλου αυτού. Η οργάνωσή μου ε, διοργάνωσε μια συνεδρίαση στον ΟΗΕ με ανθρώπους που συνέβαλαν στη σύνταξη αυτού του πρωτοκόλου, καθώς και χώρες που έχουν επικυρώσει το συγκεκριμένο το πρωτόκολλο και ε, εκπρόσωποι της Επιτροπής που ήταν και οι ίδιοι παλαιότερα ε, βουλευτές. Παράδειγμά μας είναι η, η Μογγολία. Το 2013 η Μογγολία αποφάσισε κοινοβουλευτικά να επικυρώσει το, το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο καταργώντας έτσι θενατική ποινή. Επίσης, η Μογγολία συμμετέχει στην ε, ομάδα χωρών της οργάνωσής μου και πρέπει να πω ότι η οργάνωσή μου συνέβαλε μεταξύ άλλων στην ε, κατάργηση θενατικής ποινής ε, στην Μογγολία. Εκπρόσωπος του ICDP επισκέφτηκε τη Μογγολία, συζήτησε τα βήματα που θα χρειαστούν για την, καταδίκη, για την κατάργηση της θανατικής ποινή. Και για να σας πω και λίγο λόγια για το ICDP. Είναι μια οργάνωση που δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια, το 2010, ως πρωτοβουλία της ε, Ισπανικής κυβέρνησης με σκοπό να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελείται από 15 υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που υποστηρίζουν όλοι την ε, κατάρριση θανατικής ποινής. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πρώην βουλευτές. Έχουμε ε, προέδρου, πρώην προέδρους, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην ε, κυβερνητικούς αξιωματούχους, αξιωματούχους του ΟΗΕ, κυβερνήτες και δικαστές από, την, ε, από τις ίπα και ε, επιστήμονες. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στην ιστοσελίδα μας. Αυτό που είναι σημαντικό όμως για την οργάνωσή μας είναι ότι έχει την υποστήριξη 18 χωρών που ε, αντιπροσωπεύουν όλες τις ε, περιφέρειες του κόσμου. Τι κάνουμε. Το ICDP διοργανώνει διμερείς συναντήσεις με αξιωματούχους ε, χωρών που ε, θέλουν να αναλάβουν δράση για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Φέτος συζητήσαμε με την κυβέρνηση της ε, ΑΙΤΙΣ και αυτό που ξέρουμε είναι ότι ε, η, είναι ότι η IT θα επικυρώσει τη συνθήκη αυτή. Επίσης το ICDP διοργανώνει αποστολή το ΛΕΣ Πρόσφατα έγινε μία στον Λίβανο και ο πρόεδρος, ο κύριος Μαγιόρ, μαζί με δύο επιτρόπους, ε, συναντήθηκε με κυβερνητικούς εκπροσώπους της, ε, του Λιβάνου. Οι βουλευτές στο Λίβανο, στη συζήτηση, στη συνάντηση που έγινε, συζήτησαν το ενδεχόμενο να γίνει ένα μορατόριουμ στις ε, εκτελέσεις. Υπάρχει μια κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς παρακολουθούμε τις ε, αλλαγές. Εκτός από τις διμερείς ε, επαφές, τις ε, επισκέψεις και τη συνεργασία μας με διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΟΗΕ, το ICDP επίσης εκδίδει άρθρα. Μάλιστα, στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα εκδοθεί και ένα σχετικό βιβλίο, όπου ο κύριος Μαγιόρ, ο πρόεδρός μας, έχει συγγράψει ένα από τα άρθρα για την κατάρριξη της ε, θανατικής Στην ε, δημοσίευση αυτού του βιβλίου θα, θα παραστεί και ο κύριος Μπαν Κιμούν και εκπρόσωποι ε, χωρών ε, από όλο τον κόσμο και μεταξύ αυτών και εκπρόσωπος της Ιταλικής Κυβέρνησης. Επίσης εκδώσαμε πέρσι μια έκθεση για το πώς οι χώρες κατάργησαν τη θανατική ποινή. Πρόκειται για μια συλλογή 13 ε, χωρών που έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή και σε όλες τις περιπτώσεις οι βουλευτές διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο για την κατάργηση. Για να επανέλθω τώρα στη συνάντηση που έγινε πέρσι με βουλευτές, είδαμε ότι έχουν συγκεκριμένο ρόλο να, να διαδραματίσουν οι βουλευτές. Για παράδειγμα, όσον αφορά την, ε, την υιοθέτηση νομοθεσίας για την κατάρριξη ποινής, αλλά και για την μείωση των ε, αδικημάτων που ε, τιμωρούνται με θάνατο. Επίσης, οι βουλευτές μπορούν να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα. Επίσης θα γίνουν συναντήσεις και επισκέψεις με βουλευτές χωρών που δραστηριοποιούνται υπέρ της καταρρήσης της θανατικής ποινής. Συναντήσαμε ε, ε βουλευτές από το Σουρινάμ, ε, και από την Καραϊβική και θα θέλαμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στο μέλλον σε αυτές τις αποστολές. Σε αυτές τις επισκέψεις οι βουλευτές έχουν πάντοτε την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσουν αυτά που θα μάθουν στον τύπο. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε και πολλές προκλήσεις. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με τον ΟΗΕ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους συναδέλφους από την ε, ε, Διεθνή Αμνηστία, τη Ριμπρίφ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως υπόθηκε, το κίνημα κατά της θανατικής ποινής γίνεται όλο και ισχυρότερο. 153 χώρες έχουν καταργήσει θανατική ποινή ή δεν εκτελούν ανθρώπους. Αλλά υπάρχουν ε, και προβλήματα. Για παράδειγμα, Αίγυπτος, Νιγηρία, Σιγκαπούρη, ε, η Δονησία, Κουβέιτ φέτος έχουν ε, επαναφέρει την ε, θανατική ποινή. Επίσης, ε, στην Ευρώπη, στη Λευκορωσία εξακολουθούν να γίνονται εκτελέσεις. Έχουμε την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, που, όπου γίνονται πολλές εκτελέσεις και έχουμε και μαζικές δίκες στην Αίγυπτο, οι οποίες κατέληξαν ε, το Μάρτι και ε, τον Απρίλιο 1.200 ε, άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο σε μία δίκη από έναν δικαστή. Επίσης υπάρχουν κινήσεις στο Μάλι, στο Μπρουνέι, στην Ιγυρία για την, για την διεύρυνση της χρήσης της θανατικής ποινής. Είχαμε και ε, εκτελέσεις στην Αριζόνα και στην Οκλαχώμα φέτος οι οποίες δεν εκτελέστηκαν ε, με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Τον Απρίλιο ο Έπλη Λόκετ από την Οκλαχώμα η εκτέλεσή του διήρκησε πάνω από 43 λεπτά. Τον Ιούλιο στην Αριζόνα εκτέλεση με θανατηφόρα ένση διήρκησε 177 λεπτά. Επίσης να επισημάνω ότι τον Ιούλιο για πρώτη φορά ένας δικαστής της Καλιφόρνιας είπε ότι η θανατική ποινή είναι αντισυνταγματική διότι έρχεται σε αντίθεση με την 8η τροπολογία του συντάγματος των ήπα που απαγορεύει την ε, απάνθρωπη μεταχείριση, μετα, ε, μεταχείριση ανθρώπων. Και θα ήθελα να τελειώσω ε, αναφέροντας αυτό που λέει ο κύριος Μαγιόρ. Η απόρριψη της ε, θεανατικής ποινής περιλαμβάνει το τι ε, κοινωνία θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε σε μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία. Και γι' αυτό καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει τον ε, ρόλο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόμαστε σε επαφή ε, με βουλευτές από όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε ότι θα καταργηθεί σε όλο τον κόσμο η θανατική ποινή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ντέβιτ Νίκλας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας καλήσατε, καλέσατε εδώ για να μιλήσουμε επ' ευκαιρία της ε, Παγκόσμιας ημέρας κατά της θανατικής ποινής στη 10η Οκτωβρίου. Πράγματι εστιάζουμε φέτος στη χρήση της θανατικής ποινής ε, κατά ανθρώπων που έχουν ψυχική ε, νοητική αναπηρία παρά το ότι τα διεθνή πρότυπα λένε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται σε τέτοια άτομα η θανατική ποινή, αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει σε πολλές χώρες. Να σας δώσω παραδείγματα από φέτο από τι ΗΠΑ τον Ιανουάριο, ο Αστούραλ Μαχάμετ εκτελέστηκε στην ε, Φλόριντα παρότι είχε ένα μακρό ιστορικό σοβαρής ψυχικής ασθένειας. Ε, ήταν ε, συγκεκριμένα έπασχε από παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Αυτόν Απρίλιο ένας Μεξικανός και ο Φερνάντες Λάμας, εκτελέστηκε στο Τέξας παρά τα αποτελέσματα δοκιμών και τα στοιχεία που έδειχναν ότι είχε νοητική αναπηρία και περιμένουμε τώρα ε, πάρα πολλοί ε, άνθρωποι ε, τη θέσηρά τους για εκτέλεση, ενώ πάσχουν από σοβαρά νοητικά ή ψυχικά προβλήματα. Ανέφερε προλαλή το πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή θανατική ποινή, έδωσε κάποια στοιχεία. Σίγουρα υπάρχει μια τάση παγκόσμια για την κατάργηση. Υπάρχουν λίγες ε, ε, χώρες που εκτελούν ανθρώπους, λιγότερες από ό,τι παλιότερα και όσες εκτελούν ανθρώπους ε, απομονώνονται. 22 χώρες, 22 εκτελέσεις μάλλον είχαμε το 2013 και βλέπουμε ότι κυρίως στην Αφρική υπάρχει ηγετική συμπεριφορά από πολλές ε, κυβερνήσεις που αναθεωρούν την νομοθεσία τους για τη θανατική ποινή. Παρ' αυτά το 2013 αλλά και μέχρι τώρα το 2014 βλέπουμε αρνητικές τάσεις και ανησυχητικά μηνύματα λαμβάνουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε εκτελέσεις και πάλι στην Ευρώπη όπως αναφέρθηκε με τουλάχιστον δύο εκτελέσεις στη Λευκορωσία υπό συνθήκες πλήρους μυστικότητας τον Απρίλιο. Δεύτερο είδαμε ε, ξανά εκτελέσει σε πολλές χώρες ε, που de facto Υπήρχε μορατόριο όπως ε, Νιγηρία, Βιετνάμ και άλλες χώρες που αναφέρθηκαν και σε αυτές τις χώρες οι εκτελέσεις σε μεγάλο βαθμό έγιναν πάλι σχεδόν σε άκρα μυστικότητα. Τρίτον, έχουμε δει αύξηση των εκτελέσεων μικρότερες χώρες αλλά που εκτελούν περισσότερους ανθρώπους. Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον 59 εκτελέσει είχαμε με, μέχρι τώρα το 2014. Είδαμε επίσης στη Σαουδική Αραβία την εκτέλεση ανθρώπων ε, που υποτίθεται ότι διάπραξαν τα εγκλήματά τους σε ηλικία κάτω των 16 ετών. Αυτό παραβιάζει τη διεθνή νομοθεσία, η εκτέλεση δηλαδή. Επίσης στο Ιράκ έχουμε κάθε χρόνο αύξηση των εκτελέσεων. Οι περισσότερες γίνονται με τη χρήση ασαφών ε, αντιτρομοκρατικών ε, διατάξεων 369 ε, ήταν οι εκτελέσει που καταγράφηκαν στο ΕΡΑΝ το 2013, αλλά μάλλον υπερβαίνουν του 700 αυτοί που πραγματικά εκτελέστηκαν. Περνάμε τώρα από αυτή τη μάλλον ζωφερή εικόνα σε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό που μπορεί να κάνουν ε, τα μέλη τη υποεπιτροπή σα. Υπάρχουν ε, αρκετά πρακτικά μέτρα και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποινή, νομίζω ότι μπορούν και τα κράτη-μέλη ε, και ε, οι συνάδελφοι σας από την Υποεπιτροπή να τα προωθήσουν. Θα σας Αναφέρω ορισμένα. Πρώτα απ' όλα, κατάσταση των χωρών συγκεκριμένα. Η θανατική ποινή πρέπει να τίθεται συγκεκριμένα ε, στις χώρες και στις κυβερνήσεις ε, ε, που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική όταν έρχονται είτε εκπρόσωποι εδώ είτε πηγαίνουν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες εκεί. Και θα πρέπει να τίθεται το ίδιο θέμα και σε αξιωματούχους που έρχονται από τρίτες χώρες. Επειδή επίση αναφέρθηκε για τη ε, συνάδελφό μου, οι κοινοβουλευτικέ επαφέ είναι κάτι που δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Έχει μεγάλη σημασία. Οι κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείε του Κοινοβουλίου ε, που μιλούν για την κατάργηση τη θανατική ποινή ε, στου βουλευτέ αυτών των χωρών έδειξε ότι κάνει τη διαφορά. Και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην ενεργοποίηση μορατόριου ε, θα πρέπει όμως να υπάρξουν και προσωρινά μέτρα για την μείωση των εκτελέσεων ή την απόδοση της αντικής ποινής. Παραδείγματος χάρη να υπάρχουν περιορισμοί για ηλικιωμένους, ανήλικους, άτομα με νοητική ψυχική νόσο, να μην εκτελούνται τέτοια άτομα. Τουλάχιστον αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τώρα, τι μπορεί να γίνει. Ε, έχουν ήδη γίνει πολλά, μπορούν να μειωθούν ε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, ανθρώπους ε, υπό εκτέλεση, υπό ε, είναι σε κίνδυνο εκτέλεση. Πολλοί συνηθίζουν σε πολλέ χώρε αυτό να το κάνουν ε, όσο το δυνατόν πιο μυστικά γίνεται. Ε, άρα εμεί πρέπει να φροντίσουμε να γίνεται ντόρο για κάθε τέτοια περίπτωση. Μπορούν δηλαδή οι βουλευτέ ε, να δημοσιοποιούν τα στοιχεία, να αναφέρουν ε, τα θέματα αυτά στα δικτύα τα κοινωνικά, να ζητούν να μιλήσουν με του πρέσβει, με τι αρχέ, να κάνουν επίσημα διαβήματα. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, ε, η παρέμβαση σε υψηλό επίπεδο είναι απαραίτητη για να σταματήσει μια εκτέλεση, να ανασταλεί μια εκτέλεση. Θα μπορούσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να κάνει μια παρέμβαση στους ε, υπουργούς εξωτερικών ε, της ΕΕ ή στην ΥΠΑΤΙΚ πρόσωπο όταν αναλάβει τα αξιώματά της, να μην περιμένει μετά την εκτέλεση για να εκδώσει μια καταδικαστική ανακοίνωση, αλλά να δράει τον προτέρων. Αυτό έχει αποδώσει το παρελθόν, έχει σταματήσει εκτελέσεις. Τρίτον, μπορεί να γίνει κάτι και για την στήριξη της διεθνούς δράσης. Έχουμε το πέμπτο ψήφισμα για μορατόριο της αντικής ποινής στο πλαίσιο του ΟΗΕ και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη σε αυτό το κίνημα κατά της θανατικής ποινής ανά τον κόσμο και θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις χώρες να υιοθετήσουν μορατόριο ε, κατάργηση θανατικής ποινής. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι θέμα ποινική δικαιοσύνης θανατική ποινή. Επίσης είναι σημαντικό να δείξουμε ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη παγκόσμια τάση προς την κατάργηση της θανατικής ποινής. Αυτό πρέπει να προβληθεί. Και ε, από αυτό το πρίσμα πρέπει να κάνουμε πάντο δυνατό για να ενθαρρύνουμε περισσότερες χώρες να στηρίξουν ε, και να συνυπογράψουν το ψήφισμα του φθινοπόρου, να ενθαρρύνουν τις χώρες που έχουν θεατική ποινή να απόσχουν από την τελική ψηφοφορία και να μην υπογράψουν ε, δηλώσεις ε, διαφοροποίησης. Και σε ό,τι αφορά το κείμενο του ψηφίσματος θα πρέπει να φροντίσουμε να μην αποδυναμωθεί σε σχέση με το κείμενο του 2012. Τέλος, θα ήθελα να θέσω το ζήτημα του κανονισμού για τα βασανιστήρια είναι ένας κανονισμός που επανέρχεται στο Κοινοβούλιο. Εγκρίθηκε το 2005. Ήταν ένας πολύ σημαντικός κανονισμός. Βοήθησε ευρωπαϊκές εταιρείες να μην γίνονται συνένοχες, να μην στέλνουν ε, ε, εξαρτήματα, προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανισμό ή για θανατική ποινή. Υπάρχουν όμως παραθυράκια, σε τρίτες χώρες εννοούμε. Υπάρχουν παραθυράκια και αυτά τα πρέπει να τα κλείσουμε τώρα. Τρία είναι τα βασικά παραθυράκια που πρέπει να να παραλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή στον κανονισμό δεν υπάρχει έλεγχος ε, ε, στη μεσητεία, στο brokering. Δηλαδή μπορούν ε, να εμπορεύονται οι εταιρείε τέτοια αντικείμενα αρκεί να μην μπαίνουν αυτά τα αντικείμενα στο, στην επικράτεια της Ένωσης. Δεύτερον, δεν υπάρχει απαγόρευση της προώθησης του εξοπλισμού από ευρωπαϊκές εταιρείες, είτε στις ιστοσελίδες τους, είτε σε σαλόνια εμπορικά, εκθέσεις εμπορικές. Και έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή αντικείμενα τα οποία ποτέ θα έπρεπε να απαγορεύονται, να προβάλλονται και να προωθούνται σε εμπορικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, Υπάρχουν περιορισμοί στο όλο σύστημα και κυρίως στην αντίδραση σε καταστάσεις εκτακτής ανάγκης. Όταν ε, βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία δεν μπορεί να αντιδράσει γρήγορα για να αλλάξει ε, μια απόφαση και να δράσει γρήγορα, να προλάβει. Θα πρέπει λοιπόν να μπει μια σχετική ρήτρα. Το λέει και το Κοινοβούλιο με ψήφισμά το 2010. Ο κανονισμός όμως ήταν πολύ σημαντικός, κυρίως ε, αποτρέποντας τη συνενοχή, όπως είπαμε, για την ε, χρήση ε, φαρμάκων για την εκτέλεση μελοθανάτων από τη ΣΥΠΑ ή αλλού. Και αυτά είχα να πω. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Thank you, David Nichols. Σε ευχαριστούμε κύριε Νίκολς ε, και τώρα η Μάγια Φώ για τις αντιφόρες αυτές ε, ενέσεις και τον εμπορικό έλεγχο φαρμάκων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατικές εκτελέσεις. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια sites που επισκέπτομαι πολύ και το ένα είναι που είναι το κέντρο ενημέρωσης για τη θανατική ποινή και τις επερχόμενες εκτελέσεις. Πολλά ζωφερά στοιχεία, αλλά και ελπίδες τελευταία, γιατί αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι πολύ περιορισμένος αριθμός ε, πολιτιών στη ΣΥΠΑ που μπορούν να εκτελέσουν και γι' αυτό για τεχνικούς λόγους, γιατί δεν μπορούν να βρουν τα φάρμακα ή γιατί έχουν πρόβλημα ή γιατί δεν έχουν κατάλληλο πρωτόκολλο. Και είναι αυτό πολύ εντυπωσιακό. Την περασμένη εβδομάδα η Πενσιλβανία χρειάστηκε να αναβάλει μια εκτέλεση γιατί δεν είχε το... το φάρμακο. Η Γεωργία το ίδιο λέει ότι δεν είχαν ε, εντάλματα και μια εβδομάδα μετά μάθαμε ότι ήταν επειδή δεν είχε φάρμακα. Και αυτό σε όλες τις πολιτείες. Δεν είναι ένα φάρμακο, δεν είναι ε, ένα θέμα. Είναι μόνο ε, ότι υπάρχει θέμα με αυτά τα φάρμακα και ίσως να πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στην ιστορία για να πούμε γιατί είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Πριν από ένα-δύο χρόνια σας είχα μιλήσει πάλι γι' αυτό. Έχουμε προχωρήσει, αλλά μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουν γίνει πολλά λόγω των ε, διαφορών ε, για το φάρμακο αυτό, ε, τα φάρμακα μάλλον για τις ενέσεις, μειώθηκαν κατά το 1 πέμπτο λόγω αυτής της διαφοράς με την Ευρώπη. Και εδώ και 40 χρόνια είμαστε σε πολύ, ε, μάλλον είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 40 χρόνια. Και είναι εντυπωσιακό που αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ξεκίνησε ως μικρο, μια μικρή ελάχιστη βρετανική φιλανθρωπική ε, πράξη γιατί ανακαλύψαμε ότι οι βρετανικές φαρμακευτικές φαρμακοβιομηχανίες εξήγαν αυτό το φάρμακο. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είχαν έρθει τότε και να πούν εδώ ελάτε μπορείτε να φτιάξετε τον κανονισμό και να απαγορεύσετε τη μετακίνηση των φαρμάκων προς τις ΕΠΑ. Δεν το έκαναν, έβαλαν μόνο έλεγχο γιατί ήταν επίγον. Ο έλεγχος των εξαγωγών ε, ξεκίνησε το 2010. Και έτσι σταμάτησε η εξαγωγή του πρώτου φαρμάκου που ήταν το αρχικό φάρμακο που χρησιμοποιούνταν στο αρχικό κοκτέιλ θανάτου τα πρώτα χρόνια. Η εταιρεία προσπάθησε να πάει στην Ιταλία για να φτιάξει εκεί τα φάρμακα. Δουλέψαμε και στην Ιταλία και τώρα υπάρχουν ε, ένα άλλο κράτος όπου είναι υπέρ της κατάργησης θανατικής ποινής και εμπόδισαν αυτή την εταιρεία από το να φτιάξει την παραγωγή του φαρμάκου αυτό στην Ιταλία. Τώρα άλλαξαν πρωτόκολλα, προσπαθούν να φτιάξουν άλλα φάρμακα, δεν το χρησιμοποιούν πια εκείνο το πρώτο. Πάντως, ε, Πέι, Ινδί, Ισραηλινοί, δηλώνουν ότι είναι όλα ένα και πιο δύσκολο να αγοράσει κανείς αυτά τα φάρμακα τουλάχιστον από την Ευρώπη. Και θα μιλήσω για αυτούς τους ελέγχους των εξαγωγών αργότερα και το σχετικό κανονισμό, αλλά πάντως όσον αφορά την παραγωγή, είναι ενδιαφέρον ότι εδώ πολλά χρόνια λεγόταν πως οι εταιρείε δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη διανομή των φαρμάκων τους δήθεν. Ότι ήταν δηλαδή φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνταν για εκτελέσεις και ότι οι εταιρείε ήταν ανάμεσα ε, ε, ε, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ήταν μπρος και πίσω Αυτό ήταν μύθο βέβαια και οι εταιρείε μπορούν αυτό να το ελέγξουν και αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί στον ίδιο τον κανονισμό. Εμεί συναντάμε τι εταιρείε και ξεκινήσαμε με τι ευρωπαϊκέ, αλλά χρειάζεται να αναλάβουν ευθύνη για τη διανομή των φαρμάκων του, αλλά πρέπει να του βοηθήσουμε. Οπότε συνεργαζόμαστε μαζί τους για την ε, έλεγχο της διανομής των φαρμάκων, για να ε, δουλεύουμε για να δούμε πώς και πού βρίσκουν τα φάρμακα οι, οι φυλακές, να εξηγήσουμε στις εταιρείες ότι τα φάρμακά τους είναι κίνδυνος, να προστατέψουμε την ευρωπαϊκή αγορά με την αλλαγή των ε, του κανονισμού για τον έλεγχο των εξαγωγών, έτσι ώστε να μην μπορούν να βρουν τα φάρμακα να μην μπορούν να βρουν τα φάρμακα, αλλά και οι φαρμακοβιομηχανίες να προστατευτούν, γιατί δεν είναι αυτές ο εχθρός μας. Σε αυτή τη φάση λοιπόν πρέπει να εξασφαλίσουμε πώς ε, θα διαδίδονται οι καλύτερες πρακτικές σε ολόκληρη τον κλάδο, αλλά και παγκοσμίω. Ε, και αυτό που ε, ήταν πολύ σημαντικό είναι ότι είχαμε αντίκτυπο στη ΣΥΠΑ, αλλά και άμεσα και έμεσα και σε άλλες χώρες. Πάντω για την ώρα δεν μπορούσαν να εκτελέσουν γιατί δεν χρησιμοποιούν, δεν, δεν βρίσκουν τα φάρμακα και όσοι κάνουν αυτέ τι ενέσει δεν μπορούν να τις κάνουν ούτε και αυτοί γιατί ακολουθούν τη ΣΥΠΑ. Έμεσα όμω, αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι και χώρε που, άλλε που σκέφτηκαν να κάνουν τις ε, αντιφόρες ενός γιατί είναι ο πιο ανθρώπινο τρόπο για να εκτελέσουν τους ε, καταδίκου και βλέπουν τι γίνεται στη ΣΥΠΑ και το ξανασκέφτονται αν τους συμφέρει να περάσουν σε αυτό το είδος εκτέλεσης. Είναι τέτοιο τύπο που εμείς οι θεατές δεν μπορούμε να δούμε τη βιότητα της διαδικασίας. Ξέρουμε ναι, ότι είναι σε αυτό το δωμάτιο, αλλά εν γέννη για το κοινό έχει προωθηθεί, έχει παρουσιαστεί ως ανθρώπινη μέθοδος. Ψευδοϊατρική διαδικασία. Όχι, δεν είναι όμως. Και αυτό που έγινε είναι ότι στην ουσία έφυγε πια αυτό το πέπλο το ιατρικό, αυτός ο Φερετζές ο ιατρικός και έτσι φάνηκε ξεκάθαρα τι είναι. Στην Αριζόνα ξαν, πρέπει, ας πούμε, σταματήσαν τελείως οι, οι, εκτελέσεις και στην ιστορία της κατάργησης θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Το σημαντικό τώρα για τις διάφορες μεθόδους όπως ας πούμε η θάλαμη αερίων ή η ηλεκτρική καρέκλα η επιστροφή σε αυτά είναι κάτι το ελπιδοφόρο γιατί δείχνουμε ότι είναι οπισθοδρομική όλοι αυτοί άρα δεν μπορούμε να κάνουμε ε, με ανθρώπινο τρόπο τις εκτελέσεις άρα δεν έχει νόημα και να την κάνουμε δεν μπορούμε να την κάνουμε την εκτέλεση στην ουσία δεν υπάρχει ανθρώπινος τρόπος Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι θετικά. Τώρα για τους ελέγχους εξαγωγών πολύ χρήσιμα είναι τα πράγματα που υπάρχουν στον τροποποιημένο ε, κανονισμό γιατί οι εταιρείε μπορούν να συνεχίσουν να πουλάνε αυτά τα πολύ σημαντικά φάρμακα και αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν μπορεί να φανεί ότι περιορίζουμε τα φάρμακα, ότι εμποδίζουμε το εμπόριο. Οπότε να τους επιτρέψουμε να το συνεχίσουν ενώ, δίνουμε, ενώ κάνουμε πολύ πολύ αυστηρούς ελέγχους που τους αναγκάζουν και τους ενθαρρύνουν να κάνουν βήματα ώστε να ελέγξουν και εκείνοι με τη σειρά τους διανομή λειτουργεί. Έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει με εταιρείε, μπορούμε να συμβουλέψουμε, το έχουμε ήδη κάνει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τη ενθαρρύνει να το κάνουν. Είναι πολύ βοηθητικό δηλαδή το να νομοθετεί η Ευρώπη και η διαδικασία για τη τροπολογία ε, διευκόλυνε στο να προστίθενται τα φάρμακα με το που ε, ανακαλύπτονται. Έχουμε νέα πρωτόκολλα και θέλουμε να έχουμε ένα πραγματικά λειτουργικό σύστημα όπου ένα νέο φάρμακο μπορεί να φτιαχτεί, να μπει στο παράρτημα και να ελέγχεται από την Ευρώπη γρήγορα. Τώρα, πώς γίνονται όλα αυτά, πώς θα γίνουν όλα αυτά, δεν ξέρω, δεν είμαι σε αυτό το κόσμο καθημερινά, αλλά πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει γρήγορα. Και γρήγορα να κλείσω και αυτό το τμήμα της συζήτησης. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ο κύριος Αλεξανδρίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα σας ε, μιλήσω. Εξάντλησα το τέταρτο που είχα στη διάθεσή μου όταν σας μίλησα για τον Μπαχρέιν. Αλλά ήθελα να πω για την θανατική ποινή ότι είναι ένα από τα πολύ σπάνια ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινωνία των πολιτών συμβαδίζουν απόλυτα. Υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών. Δεν είμαι ποτέ καλό στα μαθηματικά. Και παρότι ε, παρακολουθώ τις στατιστικές, έχω την αίσθηση ότι φυσικά πρέπει να ε, χαρούμε για το γεγονός ότι η τάση για την κατάργηση ε, ενισχύεται, αλλά μην μας δημιουργήσει και ψεύτικες, ε, ψεύτικη αυτοπεποίθηση, διότι κάθε χρόνο είμαστε αντιμέτωποι με αρνητικές εκπλήξεις. Ο Ντέβι το είπε, πέρσι είχαμε τουλάχιστον πέντε, χρόνια, πέντε χώρες που έσπασαν πολυετή μορατόρια που υπήρχαν. Ε, χώρες που εκτέλεσαν ανθρώπους που δεν είχαν εκτελήσει από τη δεκαετία του 50 και του 60. Οι προσπάθειές μας λοιπόν πρέπει να είναι σταθερές και συστηματικές. Να τονίσω και εγώ αυτό που είπαν πολλοί ε, ομιλητές. Ε, να σας διαβεβαιώσω προσωπικά ότι ποτέ δεν υπήρξε δομημένος διάλογος με χώρα όπου ισχύει η θανατική ποινή, όπου το ζήτημα αυτό να μην τέθηκε. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες συζητήσεις, ακόμα και με στρατηγικούς εταίρους και φαντάζομαι καταλαβαίνετε σε ποιους αναφέρομαι. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, η 10η Οκτωβρίου είναι προτεραιότητα για μας. Εκτός από την ε, κλασική ε, διακήρυξη έχουμε δώσει ε, εντολή σε όλες τις αντιπροσωπείες μας, σε όλες τις χώρες, ε, ιδιαίτερα στις χώρες όπου ισχύει η θανατική ποινή, να μεταφράσουν τη διακήρυξη αυτή και να παρουσιάσουν ε, πρωτοβουλίες. Είτε πρόκειται για σεμινάρια, συνδιασκέψεις, ε, συνέδρια. Πρέπει να πω ότι η στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά μας έχει δώσει τη δυνατότητα ε, να αποκτήσουμε εικόνα και γνώση για το ποιου στόχου πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, στι ασιαστικέ χώρε αυτό που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινή γνώμη. Σε άλλε χώρε ο στόχο πρέπει να είναι μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο. Εκτό από τα κλασικά εργαλεία μα, δηλαδή δηλώσει, ανακοινώσει κτλ. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλέ φορέ. Υπάρχουν και τα τρίτη γενιά εργαλεία. Και εκεί που δίνουμε μεγάλο βάρο είναι η εκπαίδευση και δεν αναφέρομαι σε εκπαίδευση σε αξιωματούχους, αλλά σε ανθρώπους στις τρίτες χώρες, σε δικηγόρους, ε, δικαστές, ε, υπεύθυνους ε, ή φορείς λειτουργίας φυλακών. Επίσης, κατευθύνουμε χρηματοδότηση και προς αυτά τα εργαλεία νέας γενιάς και πολλές φορές ακούμε το επιχείρημα ότι η κοινή γνώμη τους ε, είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι το ερώτημα, το πρόβλημα μάλλον, δεν είναι ποιον ερωτάς, αλλά πώς διατυπώνεις το ερώτημα. Και σε αυτόν ακριβώς τον τομέα θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει η δική μας γνώση και η δική μας ε, εμπειρία. Και ε, όσον αφορά το ψήφισμα στον ΟΗΕ, έχουμε ε, αφιερώσει όλες μας τις δυνάμεις για να επιτύχει περισσότερο και από ότι το 2012. Θέλουμε περισσότερες από τις 111 ε, ψήφους. Πάντως, εμείς και απαντώ ε, και σε ορισμένα σχόλια, δεν πρόκειται να κάνουμε καμία υποχώρηση στο, όσον αφορά το κείμενο. Το κείμενο θα είναι ακόμη καλύτερο από εκείνο του 2012. Νομίζω αυτά ήθελα να πω. Σχετικά με τον ε, κανονισμό έχουμε εμπιστοσύνη στους συνομοθέτες. Ήμουν μέλος μιας μικρής επιτροπής που ξεκίνησε την αναθεώρηση των παρατημάτων και τώρα μπορώ να πω ως αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το ζήτημα πλέον έχει περάσει στα χέρια των συνομοθετών. Οπότε ε, εκείνοι είναι που πρέπει να κάνουν την δουλειά από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ κύριε Αλεξανδρίδη. Βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του θέματος, στη συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Μπορείτε να πείτε και το όνομά σας, παρακαλώ. Βεβαίως, σας ευχαριστώ. Είμαι ευρωβουλευτής, ε, τις λέγουμε από την χώρα των Βάσκων. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη θανατική ε, ποινή, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα βασανιστήρια και για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να σας μιλήσω για μια έκθεση που μπορεί να μην ε, έχετε ενημερωθεί ότι δημοσιεύτηκε στη Μαδρίτη την προηγούμενη Παρασκευή δημοσιεύτηκε και έχει εκπονηθεί από ψυχολόγους, γιατρούς, ψυχιάτρους και δύο ειδικού ηγητέ ε, των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το βασανισμό, Χουάν Μέντεθ και Μπεν Έμερσον είναι οι συντάκτε και αναλύει 45 υποθέσει ε, βασανιστήριων που κατεγράφησαν στη χώρα των Βάσκων ε, και πραγματικά ουσιαστικά επαληθεύει όλες τις ιστορίες που έχουν μελετηθεί. 15 άτομα τα οποία τα συνέλαβε η Εθνική Αστυνομία, η ε, Guardia Civil, η Πολιτοφυλακή και κάποια από την Ερτσάντσα που είναι η βασική ε, αστυνομία πέραν από... Διακόπτεται. Ναι, να μιλήσετε, αλλά να μην μακρηγορήσετε, παρακαλώ, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε διερμηνία. Only for one minute. Okay. Ε, minute. Ωραία, για ένα λεπτό αν δίνετε το λόγο. Λοιπόν, ε, τορτούρα λέγεται. Ε, και μετράει με ένα πρωτόκολλο που έχει εγκρίνει και ο ΙΕ, ε, ε Σταμούλα λέγεται, χρησιμοποιήθηκε σε μια καταδίκη 40 νέων από τη χώρα των Βάσκων, ε, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί ο δικαστής ε, δεν έδωσε δίκαιο στις μαρτυρίες και καταθέσεις των αστυνομικών. Αυτή τη στιγμή όμως οι άλλοι 28 νέοι δικάζονται στην Μαδρίτη και έχουν δώσει ανατριχιαστικές μαρτυρίες για βασανιστήρια τα οποία υπέστησαν. Επειδή μιλάμε για βασανιστήρια, πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που χρησιμοποιείται συστηματικά στη, στο βασικό, στη βασική αντιπαράθεση. Πρόεδρος. Ο κύριος Ντεμεσμάκερ θέλει επίσης το λόγο, αν θέλετε, και στα Ολλανδικά, αλλά στα Ολλανδικά. Για ένα λεπτό, ναι, ευχαριστώ. Δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε ο Σνάλφος Βάσκος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έθεσε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να υπάρχει συνέπεια εντός και εκτός και στην ε, εσωτερική και στην εξωτερική πολιτική. Δεν μπορούμε να θέλουμε να είμαστε ένα καλό παράδειγμα για τον έξω κόσμο αν μέσα στα δικά μας σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα, άρα συμφωνώ ότι πρέπει να πούμε κάτι για αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θανατική ποινή, αυτή η πρόοδος που άκουσα ότι είχε επιτελεστεί σε κάποιες χώρες ε, με παρηγορεί κάπως ε, όταν έχουμε μια τόσο σοφερή όμως παγκόσμια εικόνα και δούμε τα ποσοστά των εκτελέσεων και το γεγονός ότι είναι επικεντρωμένα σε ένα μικρό ρυθμό χωρών, αναφέρθηκε το Ιράν, ε, παράδειγμα, εκεί είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση γιατί μιλάμε για εκατοντάδες εκτελέσεις. Πραγματικά, αν το δει κανείς παραπάνω, ε, παραπάνω από μια εκτέλεση την ημέρα εκεί. Σε κάποιες χώρες προβλέπεται θανατική ποινή και για ε, το σεξουαλικό προσανατολισμό κάποιου. Διερωτώ με, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις χώρες αυτές που βάζουν ε, ε, τόσο κόσμο, που εκτελούν τόσο κόσμο. Εφαρμόζεται εντατικά σε κάποιες χώρες θανατική ποινή. Συμφωνώ και εγώ με τους ε, συναδέλφους που μίλησαν πριν από εμένα ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολεί σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω την δική μας επιτροπή. Πρέπει να αφιερώσουν πολλέ προσπάθειες στην καταπολέμηση αυτή, αυτού του φαινομένου. Και για την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού που αναφέρατε, νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Για να συμπληρωθούν τα κενά και να κλείσουν τα παραθυράκια που είπατε αυτό είναι ο στόχο μα για το άμεσο μέλλον. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να εργαστούμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Πρόεδρο, Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Νομίζω ότι έχουμε ε, εμπλουτίσει τις γνώσεις μας και τα επιχειρήματα που είχαμε στη διάθεσή μα, Αν έλθει κάποιο να μας μιλήσει πέσει αντική ποινή και κυρίω αυτά που είπε η κυρία Φώα στο γερμανικό τύπο ε, αυτή η πάρα πολύ ε, φρικτή εκτέλεση ε, που δεν πέθανε ε, αμέσως το άτομο έγινε, υπήρξε μεγάλη κατακραυγή και δεν ξέρω που ήταν στο Μιζούρι νομίζω. Είχανε το υλικό για να τον σκοτώσουν γρήγορα. Και με ρώτησε ένας δημοσιογράφος μήπως νιώθετε και δεν πρέπει να νιώθετε και εσείς υπεύθυνοι. Θα μπορούσα να σταματήσετε. Και λέω λυπούμε πολύ αλλά ο λόγος ήταν ότι αυτή η κυβέρνηση του Μιζούρι επέλεξε να χρησιμοποιήσει φάρμακα που δεν τα είχε δοκιμάσει. Δεν είχαν δοκιμαστεί σε ανθρώπου, αλλά σε ζώα μόνο. Πάντως θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτό που είπατε και ιδίω να σταματήσουμε αυτέ τι εξαγωγέ. Δεν έχει να κάνει μόνο με τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και άλλε χώρε. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτε στα διάφορα, οπότε μπορούμε να κλείσουμε.